Αγαπητοί συνάδελφοι, μπορούμε νομίζω να ξεκινήσουμε τη συνεδρίασή μας, διότι θα χρειαστεί να αφιερώσουμε πολύ χρόνο στις ψηφοφορίες. Ξεκινάμε λοιπόν ευθύ αμέσω με το πρώτο σημείο στη μερίσια διάταξη. Ψηφίζουμε δηλαδή για τους γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς να δώσω το λόγο στην κυρία Ρή, στην συγγητριά μας. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα είμαι πολύ σύντομη. Ήδη έχει γίνει μια πολύ σημαντική εργασία. Μέχρι στιγμής έχουμε 316 τροπολογίες τις οποίες πρέπει να ψηφίσουμε. Θα ήθελα καταρχάς να ευχαριστήσω και εσάς και όλους τους κοιόδης συζητητές καθώς επίσης και όλους τους συναδέλφους θεωρώ ότι μολονότι υπήρχαν αποκλήσεις απόψεων, πολλές αποκλήσεις απόψεων πολιτικές, περιφερειακές, εθνικές καταφέραμε να συσπυρώσουμε τις διάφορες απόψεις προκειμένου να καταλήξουμε σε έναν συμβιβασμό. Θεωρώ λοιπόν ότι θα καταφέρουμε να περάσουμε γρήγορα και αρμονικά στον τριμερή διάλογο. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστούμε και εμείς. Νομίζω ότι μπορούμε να ξεκινήσουμε λοιπόν με την ψηφοφορία. Έχετε το κατάλογο ψηφοφορίας όλοι. Έχετε όλοι επίσης τις κάρτες ψηφοφορίας. Πολύ ωραία. Ξεκινάμε με την τροπολογία 156 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 157 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 158 υπέρ κατά αποχές Ας ελέγξουμε ηλεκτρονική επαλήθευση. Άρτη ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 159. Έχουμε προφορική τροπολογία εδώ. Ο κύριος Στάις έχει το λόγο. Δεν υπάρχει λόγος να πάρει το λόγο. Γράφετε εδώ πέρα προφορική τροπολογία στο κείμενό σας. Υπάρχει κάποια αντίρρηση. Όχι. Ψηφίζουμε λοιπόν την τροπολογία 159 με την προφορική τροπολογία. Υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Ηλεκτρονική επαλήθευση μάλλον. Άρτη ψηφοφορία. Οι σοσιαλιστές έχουν δύο επιπλέον ψήφους, βλέπω. Συγγνώμη, Ματίας. Μία. Είμαστε εντάξει. Πέρας. Απορρίπτεται. Λυπάμαι. Συμβαστική τροπολογία υπαριθμών 1. Υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία υπαριθμών 6. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία υπαριθμών 7. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Περνάμε στη σελίδα 15 του κατάλογου ψηφοφορίας. Συγγνώμη. Συγγνώμη, δεν έχετε όλοι μάλλον την ίδια ρύθμιση. Τροπολογία 244. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 246 υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 250 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 247 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 249 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 251 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 248. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 253. Υπέρ. Σας δω συγγνώμη, 253 καταπίπτει. Περνάμε στροπολογία 252 υπέρ κατά Νομίζω ότι απορρίπτεται, αλλά στο ελέγξουμε. Άρτη ψηφοφορία. Οι σοσιαλιστές πάλι έχουν μία επιπλέον ψήφο, βλέπω. Είμαστε εντάξει, ωραία. Πέρας. Απορρίπτεται. 256. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Ας ελέγξουμε όμως ηλεκτρονικά. Πέρας. Εγκρίνεται. Σας το συγγνώμη. Εγκρίνεται. Τροπολογία 254. Υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 255. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 261 αυτή καταπίπτει. Περνάμε στην τροπολογία 25 και 256 μαζί γιατί είναι ταυτόσιμες. Υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές εγκρίνονται. Τροπολογία 257 για τη 258 καταπίπτει. Ψηφίζουμε τη 257 λοιπόν υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. ...259 της κυρίας Γκερλίν υπέρ... ...κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 262 υπέρ παρακαλώ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 26 και 263 είναι ταυτόσιμες, υπέρ παρακαλώ και για τις δύο, κατά αποχές εγκρίνονται. Θέλετε να κάνουμε ηλεκτρονική επαλήθευση. Λοιπόν, να σε επαληθεύσουμε ηλεκτρονικά για τις ε, τροπολογίες 26 και 263 παρακαλώ. η ψηφοφορία. Άρχεται η ψηφοφορία και έχουμε μία επιπλέον ψήφο πάντα από τους σοσιαλιστές. Είμαστε εντάξει τώρα. Πέρας. Εγκρίνονται. Τροπολογία 264 υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές. Δεν σηκώστε τα χέρια σας, συγγνώμη. Λοιπόν, ψηφίζουμε τη 264. Υπέρ παρακαλώ. Μα σύμφωνα με το κατάλογο ψηφοφορία μας το κάναμε. Έχετε δίκιο. Περνάμε λοιπόν στην 269. Η 267 καταπίπτει, διότι μία από τις τρεις τροπολογίες που βλέπετε εδώ πέρα στον κατάλογο ψηφοφορίας έχει εγκριθεί. Άρα ψηφίζουμε την 269. Συμφωνεί. Σε δύο τμήματα λοιπόν. Το πρώτο τμήμα, υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Ψηφίζουμε το δεύτερο τμήμα της 269 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 270 και 271 οι επόμενες τροπολογίες είναι ταυτόσιμες, αλλά καταπίπτουν διότι υπερψηφίσαμε τη 269. Συνεπώς περνάμε στην τροπολογία 273 του κ. Στάις. Υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 274. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 275. Υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Οι 28 και 277 είναι ταυτόσιμες από κοινού υπέρ παρακαλώ. αποχές εγκρίνονται. ...281 υπέρ κατά αποχές ηλεκτρονική επαλήθευση για τη 281 Πάλι μία επιπλέον ψήφος από τους σελιστές. Πέρας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 286. Υπέρ παρακαλώ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 288 σε δύο τμήματα. Ψηφίζουμε το πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα της 288 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Από κοινού τις 29 και 287. Είναι ταυτόσημες, υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές εγκρίνονται. Η 284 καταπίπτει και περνάμε στη 289. Υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές ηλεκτρονική επαλήθευση για τη 289. Άρτη ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. «290. Υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 291 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 292 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 294 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Η 296 καταπίπτει, άρα περνάμε στην τροπολογία 297. Υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Νομίζω ότι οι περισσότεροι ήταν κατάλα θα κάνουν ηλεκτρονική επαλήθευση για τη 297 άρθρη ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 298 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 31. Εφήσουμε τροπολογία 31 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 299 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Περνάμε στην τροπολογία 301 της κυρίας Σόμερ σε δύο τμήματα. Ψηφίζουμε το πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Δεύτερο τμήμα της 301 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 303 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 302 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική τροπολογία υπαριθμών 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 310 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 311 υπέρ κατά αποχές Εγκρίνεται, αλλά θα κάνουμε ηλεκτρονική επαλήθευση για αυτή την τροπολογία. 311. Άρτη ψηφοφορία. Πήσατε όλοι. Πέρας. Εγκρίνεται. Τρακόσια δώδεκα με προφορική τροπολογία του κυρίου Στάις. Υπάρχουν αντιρρήσεις για αυτή την προφορική τροπολογία. Όχι, συνεπώς ψηφίζουμε την τροπολογία 312 όπως τροποποιήθηκε με την προφορική τροπολογία υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές. Ηλεκτρονική επαλήθευση για την 312. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Εγκρίνεται. Περνάμε στις αιτιολογικές αναφορές. Τροπολογία παριθμών 1 της ηγήτριας υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία υπαριθμών 2. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Περνάμε στην τροπολογία 47 των Φλάνναγκαν και Φερέιρα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 50 σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. κατά αποχές. Νομίζω ότι εγκρίνεται, αλλά στο ελέγξουμε και ηλεκτρονικά. Μόνο για το δεύτερο τμήμα της 50. Άρτη ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 53. Υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 54 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 49 υπέρ κατά αποχές νομίζω ότι εγκρίνεται αλλά στο ελέγξουμε ηλεκτρονικά Πέρας. Απορρίπτεται. Σωστό λοιπόν που κάναμε την ηλεκτρονική επαλήθευση. Τροπολογία 52. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Νομίζω ότι απορρίπτεται, αλλά στο ελέγξουμε ηλεκτρονικά. Πέρας. Και όμως συγκρίνεται. Συγχαρητήρια. Τροπολογία 4. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 58 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται τροπολογία 57 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται συμβαστική τροπολογία υπαριθμών 4 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Τροπολογία 64. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 66. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 67. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Ηλεκτρονική επαλήθευση για την 67. Ψήφισατε όλοι. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 65. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 6 της συγγήτριας υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Ψηφίσουμε τροπολογία 72. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Votiamo adesso l'emendamento 76. Τροπολογία 76. Όλες οι προηγούμενες καταπίπτουν. αλλά δεν θα ψηφίσουμε ούτε την 76 γιατί καταπίπτουν οι 302 και 303. Περνάμε λοιπόν αμέσως στη συμβαστική τροπολογία 5. Συγγνώμη, δεν είναι πολύ εύκολο να καταλάβει κανείς αυτό το κατάλογο ψηφοφορίας. Πάντως περνάμε τώρα συμβαστική 5, υπέρ παρακαλώ, κατά. Εγκρίνεται. Τροπολογία 84, Πέτερλε. Υπέρ παρακαλώ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 110. Όσον αφορά την τολογική σκέψη 10α, Υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 119 του κυρίου Καπούτο. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Από κοινού τις 15 και 120 που είναι ταυτόσιμες. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνονται. Τροπολογία. Τροπολογία 123. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 125 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 126 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 129 υπέρ κατά, αποχές, απορρίπτεται. Από κοινού τις τροπολογίες 17 και 128 είναι ταυτόσιμες, υπέρ παρακαλώ, κατά, αποχές, εγκρίνονται. Από κοινού τις τροπολογίες 127 και 130 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνονται. Τροπολογία 131 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 132 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Ψηφίζουμε την τροπολογία 133 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 134 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 135 σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα, υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Δεν μπορούμε να ψηφίσουμε το δεύτερο τμήμα της 135. Συνεπώς περνάμε στην τροπολογία 18. Τροπολογία 18 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 19. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Περνάμε στην τροπολογία 141. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Νομίζω ότι εγκρίνεται, αλλά στο ελέγξουμε και ηλεκτρονικά. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Όντως εγκρίνεται. Περνάμε στην τροπολογία 143. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 142. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 145 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 144 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 147 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται Τροπολογία 148. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 149. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 151. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 152 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. εγκρίναμε την 312, άρα ψηφίζουμε την 154. Υπέρ παρακαλώ. Κατά. Είστε υπέρ ή κατά οι σοσιαλιστές. Υπέρ, υπέρ. Εγκρίνεται λοιπόν. Λοιπόν, ηλεκτρονική επαλήθευση ίσως είναι καλύτερα, ναι. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Απορρίπτεται. Μάλιστα. Ψηφίζουμε τώρα ηλεκτρονικά το σύνολο του σχεδίου σύστασης για δεύτερη ανάγνωση όπως τροποποιήθηκε, άρτη ψηφοφορία. Ναι, είμαστε στην τελική ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Πρέπει τώρα να αποφασίσουμε αν θα ξεκινήσουμε τις διαπραγματεύσεις. Ψηφίζουμε και γι' αυτό. Άρτη ψηφοφορία. Υπάρχει πρόβλημα με τη διερμηνία. Λοιπόν, ψηφίζουμε τώρα την απόφαση έναρξη πραγματεύσεων. Με ηλεκτρονική ψηφοφορία, παρακαλώ. Άρτη ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Σας ευχαριστώ πολύ. Και να ευχαριστήσω επίσης και την εισηγήτρια για την εξαιρετική εργασία που έκανα. Only one minute of suspension for... Να διακόψουμε για ένα λεπτό για να επιτρέψουμε στον κύριο Επίτροπο να προσέλθει. Αγαπητοί συνάδελφοι, αγαπητοί συνάδελφοι, περιμένουμε τον κύριο Επίτροπο στις 10. Οπότε έχουμε 10 λεπτά διακοπή. Cari colleghi. Αγαπητοί συνάδελφοι, είναι ιδιαίτερη ευχαρίστηση να έχουμε εδώ στην Επιτροπή μας και στην αρχή της νέας του θητείας τον Επίτροπο Μιγγέλα Αρίας Κανιέτε, Επίτροπο Αρμόδιο για τη δράση για το κλίμα και την ενέργεια, ο οποίος μας τιμά σήμερα με την παρουσία του εδώ διότι θα καταφέρουμε να έχουμε μαζί του μια πρώτη ανταλλαγή απόψεων εν ώψη των πολύ σημαντικών θεμάτων που μας περιμένουν, που θα πρέπει εμείς εδώ στην Επιτροπή μας να αντιμετωπίσουμε τους επόμενους μήνες, αλλά και υπό το φως των διαπραγματεύσεων όσον αφορά την πολιτική κλιματικών αλλαγών πολιτική που θα μας απασχολήσει και τον Δεκέμβριο με τη διάσκεψη των ΟΕΕ για την κλιματική αλλαγή στην Λίμα του Περού και ελπίζουμε ότι θα καταφέρουμε στη συνέχεια να καταλήξουμε σε μια παγκόσμια συμφωνία στη διάσκεψη των Παρισίων το 2015. Οι νομοθετικές προτάσεις τις οποίες επεξεργαζόμαστε στην Επιτραπή μας και που έχουν να κάνουν με την αρμοδιότητα του Επιτρόπου είναι πάρα πολλές θα μπορούσα να αναφερθώ στο σύστημα εμπορίας εκπομπών, ETS, στην έμεση αλλαγή της χρήσης γης του ILUC. Θα μπορούσα επίσης να αναφερθώ στις εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα, καθώς επίσης και στις ε, τροποποιήσεις ε, που θα γίνουν όσον αφορά το πρωτόκολλο. Όλα αυτά τα ζητήματα θα μας απασχολήσουν τους επόμενους μήνες με τον Επίτροπο και ως ε, Επιτροπή Περιβάλλοντος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα έχουμε μια ηγετική θέση για τους επόμενους μήνες και τα επόμενα χρόνια. Χαίρομαι ιδιαίτερα λοιπόν που έχουμε μαζί μας τον Επίτροπο Μιγκέλα Αρία Σκανιέτη για να μας μιλήσει για όλα αυτά τα ζητήματα. Θα του δώσω ευθύ αμέσω το λόγο για να μας κάνει την παρουσίασή του και στη συνέχεια θα έχουμε τη δυνατότητα να υποβάλουμε πολλές ερωτήσεις τις οποίες σίγουρα θα μας απαντήσει ο Επίτροπος. Δίνω λοιπόν ευθύ αμέσω το λόγο στον Επίτροπο Μιγγέλα Ρία Κανιέτε. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί Ευρωβουλευτέ. Καταρχά, να ξεκινήσω την πρώτη ομιλία μου ω Επίτροπο ενώπιον τη Επιτροπή ΕΝΒΗ, τονίζοντα, όπω έκανα και κατά την ακρόασή μου, τη σημασία που αποδίδω στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όχι μόνο ως συνομοθέτη, αλλά επίση ε, στο θεσμό που με τον πιο άμεσο τρόπο εκπροσωπεί την Ευρωπαϊκή Δημοκρατία. Γι' αυτό το λόγο αποφάσισα η πρώτη μου δημόσια παρέμβαση ως Επιτρόπου να είναι ενώπιον σας σήμερα. Κατά την ακρόασή μου υποσχέθηκα ότι θα έχω ανοιχτό και διαφανή πολιτικό διάλογο μαζί σας. Για μένα αυτή η πρώτη ανταλλαγή απόψεων είναι το πρώτο βήμα στην ε, ε, ενίσχυση αυτού του διαλόγου. Ο διάλογος αυτός πρέπει να είναι ένας από τους πυλώνες για να επιτύχουμε την, ε, κλιματική, ε, την πολιτική κλιματικής αλλαγής που ε, θέλει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Αγαπητοί Ευρωβουλευτές, το κλίμα αλλάζει και τα αποτελέσματα είναι όλο και πιο καθημερινά για τους πολίτες, τις επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά. Τα επιστημονικά απορίσματα του IPCC είναι σαφή όσον αφορά το θέμα αυτό, αλλά μας δίνουν επίσης και ένα μήνυμα ελπίδας, όπως υπογραμμίζει η πέμπτη έκθεση αποτίμησης. Το μήνυμα είναι σαφές είναι εντό των δυνάμεών μα να αντιμετωπίσουμε την κλιματική αλλαγή και να περιορίσουμε το, την υπερθέρμανση σε λιγότερο από 2 βαθμού Κελσίου. Έχουμε μια επιλογή και πρέπει να έχουμε το πολιτικό θάρρο να δράσουμε τώρα φιλόδοξα και συλλογικά. Αυτό πρέπει να είναι η κοινή πολιτική μα δέσμευση τα επόμενα χρόνια και είμαι πεπισμένο ότι θα μπορώ να βασιστώ και εσά για να καταδείξουμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση διατηρεί την ηγετική τη θέση για την κλιματική αλλαγή. Πριν από τρει εβδομάδε οι ηγέτε των χωρών μας κατέληξαν σε ιστορική συμφωνία για τους πρωταρχικού στόχους και την βασική αρχιτεκτονική της πολιτικής μας για το κλίμα και την ενέργεια για την επόμενη δεκαετία, τη λεγόμενη, το λεγόμενο πλαίσιο 2030 για το κλίμα και την ενεργειακή πολιτική. Αυτό το αποτέλεσμα είναι αυτή, το επίτευγμα είναι αποτέλεσμα κοινών προσπαθειών του Συμβουλίου, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και άλλων θεσμών και του ε, καρποφόρου διαλόγου με τους εμπλεκόμενους φορείς. Τα πορίσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου δημιούργησαν πολύ θετική ενέργεια που πρέπει να μας βοηθήσει για να προχωρήσουμε και σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο. Γι' αυτό θα ήθελε η Ευρωπαϊκή Ένωση να συνεχίσει να ε, αγωνίζεται για μια φιλόδοξη πολιτική για το κλίμα και να είναι επικεφαλής των διεθνών διαπραγματεύσεων για να υπάρξει μια δεσμευτική συμφωνία στη διάσκεψη στο Παρίσι το 2015. Πρώτα απ' όλα όμω πρέπει να εργαστούμε για να έχουμε μια σύντομη και σωστή εφαρμογή του πλαισίου για το 2030. Πρέπει να το κάνουμε με ευφυή τρόπο για να έχουμε τα πληροφέλη από αυτή τη μεταβατική περίοδο προς μια, περίοδο, οικονομία λιγότερου άνθρακα για να έχουμε δημιουργία και θέσεων εργασία και ανάπτυξη. Το πλαίσιο 2030 πρέπει να γίνει συγκεκριμένη δράση, ούτω ώστε η Ευρωπαϊκή Ένωση να παραμείνει ηγέτη ε, για τι ανανεώσιμες για περισσότερη ενεργειακή αποδοτικότητα, να αξιοποιήσουμε πλήρω το δυναμικό τη πράσινη οικονομία με τον καλύτερο τρόπο από πλευρά κόστου για τα δημόσια οικονομικά, του καταναλωτέ, ε, την βιομηχανία. Πρέπει να έχουμε συγκεκριμένα μέτρα για να εφαρμόσουμε το πλαίσιο 2030. Πριν όμω αναφερθώ σε αυτά, να πω μερικά για τι γενικέ κατευθύνσει του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Καλωσορίζω θερμά την έγκριση των δεσμευτικών στόχων για μείωση των αερίων καυσαερίου για 40% και τους υποστόχους για μείωση 43% στα πλαίσια του συστήματος εμπορίας και 30%, 30% για τους τομείς που δεν υπάγονται στο σύστημα εμπορίας. Καλωσορίζω το Ευρωπαϊκό, ότι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο συμφωνεί με τις προτάσεις της Επιτροπής για να είναι δεσμευτικός ο στόχος 27% για τις ανανεώσιμες μέχρι το 2030 στην Ευρώπη. Αυτό είναι σαφές μήνυμα προς τους επενδυτές ότι θα συνεχίσουμε να προωθούμε ισχυρή ανάπτυξη στα ανανεώσιμα και να μπορέσουμε να έχουμε μια πιο ευρωπαϊκή προσέγγιση για την ενεργειακή αποδοτικότητα. Είναι αλήθεια ότι θα επιθυμούσαμε να είχαμε πιο αισιόδοξου στόχου. Η Επιτροπή πρότεινε ένα στόχο 30%. Ο πρόεδρος Γιούνκερ και εγώ είχαμε ε, ζητήσει δεσμευτική, δεσμευτικούς και όχι απλώς ε, ενδεικτικούς στόχους. Όμως αυτή η αρχική πρόταση θα υποβληθεί σε ρήτρα αναθεώρησης. Με στόχο το 30% θα κάνουμε ό,τι μπορούμε, ούτω ώστε να έχουμε μια πιο φιλόδοξη προσέγγιση. Τονίζω ένα πολύ θετικό στοιχείο. Το 40% είναι δεσμευτικός εσωτερικός στόχος. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να επιτευχθεί στην Ένωση ούτω ώστε να μην χρησιμοποιήσουμε περαιτέρω διεθνή δικαιώματα μετά το 2020. Όλε οι επενδύσει λοιπόν πρέπει να γίνουν εντό τη Ένωση. Καλωσορίζω την αρχή ότι πρέπει να έχουμε στόχους και για τους τομείς που δεν υπάρχονται στο ETS. Οι εθνικοί στόχοι πρέπει να τεθούν μεταξύ του 0 και του μείον 40% σε σχέση με τα επίπεδα του 2005 και πρέπει να συμβάλλουν στο συλλογικό μείον 30% σε αυτούς τους τομείς σε όλη την ε, έκταση της Ένωσης. Λόγω των, των φιλόδοξων στόχων για τις μειώσεις στον ε, τομέα που δεν υπάρχει στο ETS χρειαζόμαστε μεγάλη ελαστικότητα. Πρέπει να επαγρυπνούμε στα πλαίσια αυτά να διατηρηθεί η περιβαλλοντική διάσταση του συστήματος. Καλωσορίζω δύο σημαντικά μέσα χρηματοδότηση. Πρώτον, το Ταμείο για Καινοτομία για τις Επιχειρήσεις, το λυκόμενο ΝΕΡ 400 και δεύτερον, το Ταμείο Εξχρονισμού για τα κρατη με, ε, κράτη -μέλη με το χαμηλότερο εισόδημα. Αυτό σημαίνει ότι θα έχουμε 700 εκατομμύρια δικαιώματα που θα μπορούμε να αξιοποιήσουμε για να γίνει πιο αποτελεσματική η Ένωση στους τομείς αυτούς. Καλωσορίζω θερμά τις αναφορές σε ένα σωστά λειτουργών αναθεωρημένο σύστημα εκπομπών που θα πρέπει να είναι ακρογωνιαίος λίθος της πολιτικής μας για το κλίμα. Θέλω το σύστημα αυτό να παίξει πλήρως το ρόλο του ως ε, ε, αποτελεσματικό και σε όλη, τη διάρκεια της, ε, σε όλη την επικράτεια της Ένωσης σύστημα. Ένα καλό λειτουργών τέτοιο σύστημα θα ενισχύσει τη λειτουργία τη εσωτερική αγορά ενέργεια, θα βοηθήσει για να έχουμε περισσότερε ανανεώσιμε και θα βοηθήσει επίση την αύξηση τη ε, αποδοτικότητα. Και τελευταίο αλλά πολύ σημαντικό, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο αναγνώρισε τη θεμελιώδη σημασία του εσωτερικού, της εσωτερικής αγοράς ενέργειας. Και στα πλαίσια αυτά πρέπει να επιτύχουμε χωρίς καθυστέρηση το 10% διασύνδεσης των ε, ηλεκτρικών δικτύων μέχρι το 2020 και 15% μέχρι το 2030 όπως πρότεινε η Επιτροπή. Όλοι γνωρίζουμε ότι αν επιτύχουμε αυτό το στόχο διασύνδεσης θα βελτιώσει την ενεργειακή ασφάλεια και την ε, ενοποίηση των αγορών. Επίσης θα διευκολύνει την ε, εισδοχή υψηλότερου ποσοστού ανανεώσιμων στην παραγωγή ενέργειας. Γι' αυτό πρέπει να εφαρμόσουμε κρίσιμα προγράμματα κοινού συμφέροντος. Κύριε ευρωβουλευτέ, τα στοιχεία που ανέφερα προηγουμένω μας φέρνουν στο θέμα που αντιμετωπίζετε το αποθεματικό για σταθερότητα της αγοράς. Ελπίζω η εργασία σας ε, να οδηγήσει στην έγκαιρη έγκρισή του. Οπωσδήποτε αυτό θα σταθεροποιήσει το ETS της Ένωσης και θα το κάνει πιο ανθεκτικό. Και σε αυτό, όπως και σε άλλα νομοθετήματα που προτείνει η Επιτροπή, θα κάνουμε ό,τι μπορούμε, ούτω ώστε να εφαρμοστεί η συνθήκη όσον αφορά τις αρμοδιότητες του κάθε θεσμού. Πολύ ενδιαφέροντα θέματα συζητιούνται σε σχέση με αυτό το MSR συγκεκριμένα αν θα μπορούσε να ξεκινήσει νωρίτερα και αν θα μπορούσαμε αυτά τα 900 εκατομμύρια δικαιώματα του όπιστου βαρούς προγραμματισμού να πάνε κατευθείαν στο παθηματικό. Όπως τόνισα ήδη, υπάρχει πλειοψηφία στο, εάν υπάρχει πλειοψηφία στο Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο, δεν θα είμαστε κατά. Ελπίζω η εργασία για αυτό το σημαντικό νομοθέτημα να ολοκληρωθεί στο πρώτο τρίμηνο του 2015. Αν επιτύχουμε σύντομα αποτέλεσμα για το MSA, θα έχουμε δυνατότητα να υποβάλουμε όσο να τον πιο σύντομα, αλλά με βάση συμφωνία για το θέμα αυτό, νομοθετική πρόταση για να εφαρμόσουμε τη μεταρρύθμιση του ETS μετά το 2020. Το 2020. Πρόκειται για ένα φιλόδοξο χρονοδιάγραμμα. Ωστόσο, χρωστούμε στην βιομηχανή μας, καθώς και σε όλους συμμετέχοντε στην αγορά άνθρακα, τη μέγιστη βεβαιότητα για ε, του κανόνε που θα ισχύσουν μετά το 2020 για τη διαρροή άνθρακα. Γι' αυτόν τον λόγο δεσμεύομαι να, να προχωρήσουμε γρήγορα σε μια αναθεώρηση του ETS μετά την έγκριση του αποθεματικού για τη σταθερότητα της αγοράς. Σε ό,τι αφορά τους ε, στόχους για τους τομείς εκτός ε, ETS, πρόθεσή μου είναι να ξεκινήσουμε την επόμενη χρονιά μια μελέτη εξελόγηση για ζητήματα όπως είναι η ενισχυμένη ευελιξία και η ενσωμάτωση των τομέων γης και ε, δασοκομείας στο πλαίσιο μετριασμού πολύ σύντομα και διασφαλίζοντας βέβαια την καλή ποιότητα μιας τέτοιας πρότασης. Όσον αφορά την ενεργειακή αποδοτικότητα, θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε το αίτημα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου να προτείνουμε τομεί προτεραιότητας στους οποίους μπορούν να επιτευχθούν σημαντικά ενεργειακά ωφέλη από άποψη αποδοτικότητα. Στον ε, τομέα των ανανεώσιμων πηγών ε, ε, ενέργειας θα πρέπει να προτείνουμε υποστηρικτικά μέτρα για να διασφαλίσουμε την επίτευξη του δεσμευτικού σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης στόχου του 27%. Επίσης θα πρέπει να εξετάσουμε τους τρόπους με τους οποίους μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα σύστημα διακυβέρνησης διαφανές και αξιόπιστο. Θα είναι σημαντικό να προχωρήσουμε σε εξορθολογισμό των υποχρεώσεων εκθέσεων για ζητήματα ενέργειας και κλίματος. Επίσης υπάρχει το ζήτημα της ανάπτυξης της δέσμευσης και αποθήκευσης άνθρακα. Αυτό θα είναι σημαντικό για να δημιουργηθεί μια οικονομία απαλλαγμένη από τον άνθρακα έως το 2100, όπως περιγράφεται στην τελευταία έκθεση του IPCC. Θα ήθελα επίσης να ξεκινήσουμε πριν το καλοκαίρι μια ευρεία συζήτηση για τις πολιτικές μας για τις εκπομπές και τις μειώσεις των εκπομπών στις οδικές μεταφορές και να οργανώσουμε μια συνδιάσκεψη όπου όλοι οι ε, συμμετέχοντες, οι εμπλεκόμενοι θα μπορέσουν να συνέλθουν και να ε, ανταλλάξουν απόψει για το τι έχει λειτουργήσει μέχρι στιγμή και τι μπορεί να βελτιωθεί την περίοδο μετά το 2020 και θα ήθελα και τι δικέ σα απόψει. Όπω με κάθε άλλο μέτρο πολιτική για το οποίο εγώ θα είμαι ε, υπεύθυνο, αποδίδω μεγάλη σημασία στο να ακούσω τις απόψεις όλων των εμπλεκομένων. Οι κλιματολογικέ πολιτικέ δεν πρόκειται να είναι αποτελεσματικέ αν τα οικονομικά στοιχεία δεν είναι λάθο. Γι' αυτό το λόγο ότι δεν πρέπει να χάσουμε, πιστεύω ότι δεν πρέπει να χάσουμε την ευκαιρία που μα δίνεται. Από αυτή την άποψη το πακέτο απασχόληση ανάπτυξη και επενδύσεων που θα προτείνει η Κομισιόν την επόμενη, τις επόμενες εβδομάδες θα είναι μια εξαιρετική ευκαιρία για να δείξουμε την αφοσίωσή μας στην πλευρά των επενδύσεων για το κλίμα και την ενέργεια, στις υποδομές, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και ενεργειακή απόδοση. Ήδη συνεργάζομαι με την Αντιπρόεδρο Κατάινεν και όλους τους επιτρόπους που εμπλέκονται ώστε η πολιτική αυτή να αποτελέσει ε, αναπόσπαστο τμήμα του πακέτου επενδύσεων 300 δισεκατομμυρίων που έχει προτείνει ο πρόεδρος ε, Γιούγκερ. Το πακέτο αυτό θα ε, προσθέσει και στις εργασίες για την επίτευξη μιας ενεργειακής ένωσης υπό την αιγίδα του Αντιπροέδρου Σεφτσοβιτς. Αγαπητά μέλη, Αφού σας εξήγησα τους, ε, τα σχέδιά μας για την κλιματική δράση και την ενέργεια στην Ευρώπη, θα ήθελα να ε, αναφερθώ και στις ε, διεθνείς διαπραγματεύσεις μας στο δρόμο προς μια νέα συμφωνία στην ε, Συμφωνία για το Κλίμα στο Παρίσι θα είναι ορόσημο ε, η Λίμα. Θα είναι σημαντικό. Με αυτόν τον τρόπο, για αυτόν τον λόγο, ε, φιλοδοξούμε να συνεργαστούμε με το Κοινοβούλιο και με την αντιπροσωπεία της Επιτροπής σας πριν και κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων στη Λίμα. Να διασφαλίσουμε ότι η Ευρώπη θα μιλά με μία φωνή. Η συνδιάσκεψη του κλίματο στη Λίμα θα πρέπει να αποφέρει τρία αποτελέσματα. Πρώτον, να διασφαλίσουμε ότι όλοι οι διεθνεί εταίροι μα θα προσέλθουν με, τους δικούς τους με τα δικά του σχέδια για ε, την μείωση τη εκπομπή αερίων θερμοκηπίου πριν το Μάρτιο του 2015. Μια διεθνής ε, διαδικασία πρέπει να δημιουργηθεί εν ώψη της συνέντευξης του Παρισιού για να αναλυθεί η επάρκεια και η φιλοδοξία των ε, επιμέρους ε, προσπαθειών. Μόνο έτσι μπορεί να διασφαλιστεί ότι η οριστική, οι δεσμεύσει μετριασμού στην Συμφωνία του 2015 θα είναι επαρκής για να μην, μειωθεί, για να μην αυξηθεί η παγκόσμια θερμοκρασία πάνω από 2 βαθμούς Κελσίου. Δεύτερον, θα πρέπει να κάνουμε πρόοδο ε, όσον αφορά την, τον μετριασμό των εκπομπών πριν από το 2020 για τον ίδιο στόχο, για, το, για τους δύο βαθμούς Κελσίου. Και τρίτον θα πρέπει να έχουμε μια καλή κατανόηση των στοιχείων ενός κειμένου διαπραγμάτευσης που, ε, για την ε, Συμφωνία του 2015. Για να προετοιμάσουμε την συνδιάσκεψη της Λίμας, έχω ήδη ξεκινήσει να, να συζητώ με την ε, ύπατη εκπρόσωπο και αντιπρόεδρο της Ομισιόν Φεντερίκα Μογκερίνη. Στις 5 Νοεμβρίου αποφασίσαμε ότι όλες οι πληροφορίες μας, οι διπλωματικές, θα πρέπει να κινητοποιηθούν προκειμένου... Ε, ε, στις διαπραγματεύσεις στη Λίμα η κλιματική δράση να βρίσκεται στο κέντρο των εξωτερικών μας σχέσεων. Αυτό δεν θα μπορούσε να είναι και διαφορετικά αν θέλουμε το πλαίσιο του 2030 να θέσει την Ευρωπαϊκή Ένωση ε, σε ηγετική θέση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ευθύνεται μόνο για το 10% για τις παγκόσμιες ε, εκπομπές σήμερα. Είναι όμως σημαντικό να ε, όλες οι μεγάλες και αναδυόμενες οικονομίες να προσέλθουν με δικούς τους στόχους για την μείωση έως το πρώτο τρίμηνο του 2015. Επιπλέον, τους επόμενους μήνες θα προσπαθήσουμε ε, να ε, εκδώσουμε μια ανακοίνωση σχετικά με το δικό μας όραμα για την Συμφωνία του Παρισιού και τη φύση της συλλογικής παγκόσμιας προπάθειας που απαιτείται για να αντιμετωπιστεί η κλιματική αλλαγή με τρόπο που θα αντικατοπτρίζει τις ε, τρέχουσες, τους τρέχοντες συσχετισμού πρέπει να διασφαλίσουμε ότι η κλιματική αλλαγή παραμένει μία από τις σημαντικέ μας προτεραιότητες. Στου επόμενου 13 μήνες οι προσπάθειε αυτές θα συνεχίσουν και θα αποκτήσουν μεγαλύτερη σημασία. Τους επόμενους μήνες με του άλλου επιτρόπους και με την Αντιπρόεδρο θα προσπαθήσουμε να διασφαλίσουμε η κλιματική αλλαγή να παραμείνει κορυφαία προτεραιότητα στον εξωτερικό μα διάλογο. Η δράση μας και οι συγκρίσιμες προσπάθειες από τους ε, ε, διεθνούς εταίρους μας θα αμβλύνει και τις ανησυχίες από την ευρωπαϊκή ε, βιομηχανία ότι η κλιματική μας πολιτική θα μπορούσε να δημιουργήσει υπερβολικό βάρος και να μειώσει την ανταγωνιστικότητα στις διεθνείς αγορές. Είναι ενθαρρυντικό ότι πολλές χώρες ακολουθούν το παράδειγμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αναπτύσσουν και εφαρμόζουν δικούς τους, δικές τους αγορές άνθρακα, συγκεκριμένα η Κίνα, η οποία έχει ξεκινήσει διάφορα συστήματα εμπορίας εκπομπών. Θα ήθελα να ολοκληρώσω λέγοντας ότι οι δράσεις μας ε, που σας περιέγραψα σήμερα ε, θεωρώ ότι είναι ένα ε, αναπόσπαστο τμήμα της Ενεργειακής Ένωσης. Μόνο αν αντιμετωπίσουμε, μόνο με πολιτικές για το κλίμα και την ενέργεια ε, αποτελεσματικές θα μπορέσουμε να καταλήξουμε στους στόχους μας για μια πιο πράσινη ανάπτυξη και μια πιο ανθεκτική ενεργειακά οικονομία στην Ευρώπη. Κύριε Πίτροπε, ευχαριστούμε για την εισαγωγική σας παρέμβαση. Ας ξεκινήσουμε τώρα τη συζήτηση. Καταρχάς, ας ακούσουμε κάποιες ερωτήσεις από τους συντονιστές ή τους εκπροσώπους των πολιτικών ομάδων και στη συνέχεια θα ακούσουμε τις δικές σας απαντήσεις για τα ερωτήματα αυτά κύριε Επίτροπε και στη συνέχεια θα κάνουμε ένα δεύτερο γύρο ερωτήσεων με όλους τους υπόλοιπους συναδέλφους που επιθυμούν να πάρουν το λόγο. Σας παρακαλώ πολύ. Σας ζητώ να περιορίσετε τις παρεμβάσεις σας στα δύο λεπτά, προκειμένου να έχουμε το χρόνο όλοι να πάρουμε το λόγο. Ξεκινάμε λοιπόν με το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα. Άλλη Μπέλετ, έχετε το λόγο για δύο λεπτά. Uh, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, καλημέρα σας. Και σας συγχαίρω για την ε, για το διορισμό σας. Σίγουρα είναι κρίσιμο το χαρτοφυλάκιό σας για το περιβάλλον, για την οικονομία, για τις θέσεις εργασίας. Το πακέτο για την ανάπτυξη και τις επενδύσεις και τις θέσεις εργασίας ε, είναι πολύ ζωτικό και ζωτικό τμήμα του αυτό που αφορά την κλιματική αλλαγή και την πράσινη οικονομία. Πολύ συγκεκριμένες ερωτήσεις για να τηρήσω και το χρόνο που πρότεινε ο Πρόεδρός μας. Αναφερθήκατε στα απορίσματα του Συμβουλίου πριν από 15 μέρες. Το Συμβούλιο είναι κάπως πιο μετριοπαθές ε, και το λέω και εγώ μετριοπαθώς σε σχέση με την άποψη του Κοινοβουλίου. Χαίρομαι λοιπόν που εσείς εμένετε στους στόχους σας για την ε, ενεργειακή αποδοτικότητα. Μιλήσατε για τη ρήτρα αναθεώρησης Μπορείτε να είστε πιο συγκεκριμένο, Πώς θα γίνει αυτή η αναθεώρηση. Πώς μπορούμε να προσπαθήσουμε να επιτύχουμε αυτό το στόχο του 30% για την ενεργειακή αποδοτικότητα που είναι το ελάχιστο. Δεύτερον, οι συνδιασκέψει ΚΟΠ, Λίμα, Παρίσι. Φυσικά, σας στηρίζουμε σε αυτά που είπατε. Αλλά ποιο θα ήταν ένα ελάχιστο αποτελέσμα για τη Λίμα και ιδίω για το Παρίσι. Και τι θα συμβεί εάν δεν επιτύχουμε σε κατάληξη συμφωνίας. Τι εναλλακτικό σχέδιο έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση για την μετά Παρίσι περίοδο. Και τρίτον, καλωσορίζουμε το ότι αναφερθήκατε ιδιαίτερα στην ε, μεταρρύθμιση του ETS μέσω του MSR. Είστε πολύ φιλόδοξος. Αναγγείλατε ότι θέλετε συμφωνία πριν το καλοκαίρι. Ελπίζω να προλάβετε μέσω επιτυχών διαπραγματεύσεων με το Συμβούλιο. Το κύριο όμως είναι ότι υπάρχουν πολλές ανησυχίες από τις ε, βιομηχανίες ε, τις ενεργοβόρες. Είπατε ότι θα αναλάβει πρωτοβουλίες η Κομισιόν. Πότε θα υποβάλει τις προτάσεις της όμως για την ε, διαρροή άνθρακα, τον κίνδυνο δηλαδή διαρροής άνθρακα μετά το 2020, ούτως ώστε να καταλήξουμε μια καλή σε μια καλή συμφωνία όχι μόνο με την Επιτροπή έμβια, αλλά με την ε, πλειονότητα του σώματος. Ευχαριστώ. Άιβο, SD, ο Ματίας Ευχαριστώ κύριε Επίτροπε. Ευχαριστώ που ως πρώτος Επίτροπος ήρθατε εδώ στην Επιτροπή μας που έχουμε τη δυνατότητα να συζητήσουμε μαζί σας. Το θέμα μας είναι η συνδιάσκεψη το κλίμα στο Λίμα, την οποία, η οποία θα προετοιμάσει τη συνδιάσκεψη του Παρισιού και ελπίζω και στο Συμβούλιο να γίνουν περισσότερες συζητήσεις. Εμείς εδώ ε, ε, ε εκδώσαμε ένα ψήφισμα και μάλιστα ακόμα και με την Επιτροπή Βιομηχανίας ε, ε, είχαμε αρμονικές σχέσεις και στείλαμε ένα σαφές ε, μήνυμα. Πώς θέλετε να πείσετε το Συμβούλιο ότι βρισκόμαστε δηλαδή σε μια διαδικασία η οποία μας αναγκάζει να καταλήξουμε συγκεκριμένα αποτελέσματα. Όταν κοιτώ το πώς έδρασε το Συμβούλιο και σε σχέση με το πακέτο για το κλίμα που προσπάθησε να ε, αποδυναμώσει το Κοινοβούλιο. Νομίζω ότι τα πράγματα δεν ήταν καθόλου καλά. Ε, για το MSR, ε, ο Ιβο Μπέλτ μόλις είπε αν θα τα καταφέρουμε πριν από το καλοκαίρι. Μάλλον εννοούσε του 2016-2017. ή Είπατε και στην ακρόαση σας ότι αν το Κοινοβούλιο θέλει θα μπορούσαμε να ε, ορίσουμε και μια ακόμη νωρίτερη ημερομηνία εισαγωγή του. Είπατε για τη διαρροή άνθρακα, νομίζω ότι δεν πρέπει να τα μπερδεύουμε αυτά. Την διαρροή άνθρακα με το αποθεματικό για τη σταθερότητα της αγοράς με το MSR. Νομίζω ότι πρέπει ξεχωριστά να τα εξετάσουμε αυτά τα δύο ζητήματα. Θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να ασχοληθούμε ε, με το Carbon Leakage ε, List, αν θα είναι 30 ευρώ ή 60 ευρώ. Τα νοικοκυριά πληρώνουν αυτά τα ποσά, χάνοντας έτσι από την αγοραστική τους δύναμη. Θέλετε να προχωρήσουμε σε αυτήν την διαδικασία. Ε, εγώ θα έλεγα να τα αφήσουμε και να τα δούμε ξεχωριστά, αλλά σε κάθε περίπτωση αν θέλετε να κάνετε ε, θα πρέπει να είναι πολύ καλή η πρότασή σας. Τώρα για το ETS, θέλετε σοβαρά όσον αφορά τις, ε, για, το, για, το, για τη δέσμευση και αποθήκευση άνθρακα. Θέλετε πραγματικά να, να ξεκινήσουμε αυτή τη συζήτηση. Εκεί αυτό, αυτά, γι' αυτά συζητούμε όταν δεν υπάρχουν άλλες εναλλακτικέ. Και θα κάνουμε τα πάντα ώστε αυτά τα ηλεκτροπαραγωγικά εργοστάσια να μην φύγουν από την Ευρώπη. Αλλά θέλουμε πραγματικά να δώσουμε τόσο μεγάλη σημασία και να μειώσουμε την αποτελεσματικότητα των ε, ηλεκτροπαραγωγικών εγκαταστάσεων που δεν, με μια τεχνολογία που δεν έχει ελεγχθεί ακόμη, που δεν έχει επιβεβαιωθεί επιστημονικά. Αυτό είναι ο στόχος για τα επόμενα πέντε χρόνια. Παρακαλώ πείτε μας συγκεκριμένα. E Σας ευχαριστούμε. Εξ ονόματο του ECR η κυρία Γκέρλινγκ έχει το λόγο. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε. Καλώς ήρθατε κύριε Επίτροπε. Έχω μια ερώτηση όσον αφορά το πρόγραμμα εργασίας Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ξέρω ότι συμμετέχετε στις νέες αρμοδιότητές σας για μία μόνη εβδομάδα, αλλά ξέρετε ότι εδώ πέρα στην Επιτροπή μας θέλουμε πραγματικά να δούμε ποιες ήταν οι προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής του προγράμματός σας. Και το πιο σημαντικό, μάλιστα, υπό το φως ε, της επιστολής που είδαμε από τον κύριο Τίμερμαν στις προηγούμενες αυτές ημέρες, όπου ενδεχομένως από ό,τι φαίνεται να αποσύρεται κάποια ζητήματα από το πρόγραμμα εργασίας Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Μας ενδιαφέρει σαφώς το ζήτημα της ευφύους νομοθεσίας, των ευφύους ρύθμισης, κάτι το οποίο προώθησε η προηγούμενη Επιτροπή και θα θέλαμε και εσείς να προωθήσετε το πρόγραμμα αυτό ReFit και για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, δηλαδή μια σωστή βελτιωμένη νομοθεσία για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα ήθελα να συζητήσουμε για το ζήτημα αυτό περισσότερο εδώ στην Επιτροπή μας. Λέγεται επίσης όμως στην επιστολή αυτή ότι υπάρχουν δύο ζητήματα τα οποία έχουμε ήδη εμείς αρχίσει να επεξεργαζόμαστε, τα οποία ενδεχομένω να αποσύρεται. Το πρώτο έχει να κάνει με το όλο πακέτο όσον αφορά τα ανώτατα τεχνικά όρια για τις εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα και το δεύτερο ζήτημα το οποίο επεξεργαζόμαστε πολύ είναι το νέο πακέτο, νέα δέσμη μέτρων όσον αφορά τα απορρίμματα. Τα δύο αυτά αναφέρονται σε αυτή την επιστολή ως δυνάμει ζητήματα που ενδεχομένως να αποσυρθούν από το πρόγραμμα εργασίας Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ποια είναι η δική σας η άποψη για το ζήτημα αυτό και πότε θα είστε σε θέση να μας υποβάλλετε ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα εργασίας για τους επόμενους μήνες, προκειμένου να μπορέσουμε και εμείς να εργαστούμε με βεβαιότητα. Σας ευχαριστούμε πολύ. Εξ ονόματος των Φιλελευθέρων, ο κύριος Τόμπετς έχει το λόγο. Σας ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ κύριε Επίτροπε που είστε εδώ πέρα. Μας είπατε ότι έχουμε την διάσκεψη της Λίμα το Δεκέμβριο. Θα πάτε, είπατε εσείς εκεί, θα είστε επικεφαλής της αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχετε συμφωνήσει με τον κύριο Σεφτσοβίτς ότι εσείς ουσιαστικά θα εκπροσωπείτε την Ευρωπαϊκή Ένωση σε όλες τις διεθνείς διαπραγματεύσεις, όχι μόνο στις υψηλόβαθμες συνόδους αλλά και στις κέρυες διαπραγματεύσεις που θα μας οδηγήσουν στην Σύνοδο των Παρισίων. Ουσιαστικά το δικό σας το τηλέφωνο θα δώσει η Ευρωπαϊκή Ένωση στους διάφορους συνομιλητές που θα έχουμε, τους ανθρώπους με τους, με τους οποίους διαπραγματευτούμε στις συνδιασκέψεις αυτές ή θα υπάρχει και κάποιος άλλος ε, αρμόδιος. Επίσης, το είπαν και οι συναδελφοί μου αυτό, ποιες θα είναι οι μελλοντικές ε, δεσμεύσεις ε, όσον αφορά την κλιματική αλλαγή. Υπάρχουν κάποια σημαντικά βήματα τα οποία θα πρέπει να ακολουθήσουμε, υπάρχουν κάποια ορόσημα τα οποία θα πρέπει να καλύψουμε στο δρόμο προς το Παρίσι. Σας ευχαριστούμε πολύ εξ ονόματος της Γκουε. Παρίστια Ευχαριστώ Πρόεδρε. Κύριε Κανιέτε, είπατε πολλά για να μας ε, εξηγήσετε τις, ε, τα πορίσματα του Συμβουλίου, αλλά δεν μας ε, μιλήσατε για τις δικές σας προτάσεις, μόνο ευσεβείς πόθους. Είπατε ότι υπάρχουν φιλόδοξοι στόχοι, αλλά κατά τη γνώμη μας θα μπορούσε να είναι πολύ πιο φιλόδοξη, γιατί η κλιματική αλλαγή δεν επιτρέπει αμφιβολίες και καθυστερήσεις. Χαίρομαι που άκουσα ότι η κλιματική αλλαγή είναι προφανής, γιατί δεν αποδεχόσασταν πάντα ότι αλλάζει το κλίμα, μέχρι στιγμής τουλάχιστον. Πρέπει λοιπόν να δράσουμε. Και ελπίζω να το πιστεύετε τώρα ότι αλλάζει το κλίμα. Επίση, είπατε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα συνεχίσει να είναι επικεφαλή στις διεθνή διαπραγματευσει διαπραγματεύσει Λίμα-Παρίσι. Αλλά εγώ θα έλεγα ότι δεν μιλούσε πάντα η Ένωση με μία φωνή. Αν το κάνει με μία φωνή θα είναι καινοτομία. Και όπως και προηγούμενοι είπαν, ελπίζω να μας εξηγήσετε λίγο καλύτερα πώς ακριβώς θα διεξάγετε τις διαπραγματεύσεις. Μιλήσατε για ενεργειακή αποδοτικότητα ανανεώσιμες, είπατε ότι θα υποστηρίξετε το στόχο του 27% ένα αξιόπιστο και διαφανές σύστημα διακυβέρνησης και είπατε ότι θέλετε να μειώσετε και στις μεταφορές. Αλλά ποιε είναι οι δικέ σα ιδέε, μα ζητήσατε τι δικέ μα ιδέε. Ποιε είναι οι συγκεκριμένε προτάσει σα για αυτού του στόχου που τώρα ανέφερα. Ποιε είναι οι προτάσει σα για να έχουμε μια βιώσιμη οικονομία, για θέσει απασχόληση, για να καταπολεμήσουμε ουσιαστικά την κλιματική αλλαγή. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ, λέει ο πρόεδρο. Ο κύριο Έκχαουτ για του πρασίνου. Ευχαριστώ. Καλημέρα, κύριε Επίτροπε. Χαίρομαι που μπορούμε να κάνουμε μια ανταλλαγή απόψεων επί συγκεκριμένων θεμάτων. Επαναλαμβάνω αυτό που είπε ο συνάδελφός μου Νίλ, ο φιλελεύθερος. Ξέρουμε μετά την ακρόαση ότι η Επιτροπή πάντα έλεγε ότι θα είμαστε παρόντε στι διάφορε διαπραγματεύσει για το κλίμα. Ωραίο αυτό. Αλλά το σημαντικό είναι να είναι ένα ο συνομιλητή έναντι των υπολείπων. Όχι να πάτε εσεί στη Λίμα και ίσω στο Παρίσι ο κύριο Σεύκοβι και ο κύριο μας να πάει αλλού. Ένα πρέπει να είναι πρόσωπο μα. Την επόμενη πενταετία για τι διαπραγματεύσει. Ένα θέλουμε. Δεν θέλω μια απάντηση που να λέει ναι, ναι, θα είμαστε παρόντε. Θέλω να ξέρω ποιο θα είναι παρόν. Ποιο θα είναι το πρόσωπο, ο διαπραγματευτή. Και πρέπει να είναι το ίδιο πρόσωπο. Θα θέλαμε μια σαφή απάντηση. Παρακαλώ. Τώρα για το 2030. Το πακέτο για το 2030. Τα πορίσματα του Συμβουλίου γι' αυτό. Δηλαδή, υπάρχει κάποιο πρόβλημα αν το Συμβούλιο αποφασίζει μέσω πορισμάτων, εκεί θέλει νομοφωνία. Αλλά όταν περνάμε στην νομοθεσία, είναι συνομοθεσία και για το Συμβούλιο υπάρχει η ειδική πλειοψηφία. Αλλά στο πόρισμα, στα πορίσματά του, το πρώτο, λέγεται κάτι που μας ανησυχεί. Αυτό που λένε ότι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θα ε, εξακολουθήσει να έχει υπόψη όλα τα συστήματα, όλα τα σημεία του, ε, ε, του πλαισίου για όλα τα θέματα. Αυτό θα μπορούσε να σημαίνει ότι το Συμβούλιο λέει ότι δεν μπορούμε να πειράξουμε ούτε το θέμα της ε, διασύνδεσης, ούτε το σύστημα εμπορίας, ούτε το μη εκτός εμπορίας. Πρέπει να ακολουθήσουμε αυτά που υπάρχουν στα πορίσματα. Αλλά αυτό είναι ο ελάχιστος κοινό παρονομαστής, γιατί εκεί χρειάζεται ομοφωνία του Συμβουλίου. Υπάρχουν δηλαδή 28 βέτο. Αυτό δεν ισχύει με τις νομοθετικές προτάσεις. Και κάτι που είναι σαφές ο κύριος Γιούνκερ μας υποσχέθηκε δεσμευτικούς στόχους για την ενεργειακή αποδοτικότητα. Δεσμευτικούς. Υποθέτω λοιπόν ότι το Συμβούλιο θα υποβάλει προτάσεις που να είναι δεσμευτικές. Γιατί εδώ είναι απλώς ο ελάχιστος κοινός παρονομαστής στις κατευθυντήριες. Και τελευταίο. Τα άλλα πορίσματα για τις αντισταθμίσεις, το Ταμείο Αντισταθμίσεων και η επιλογή για ε, δωρεάν δικαιώματα για αυτούς που παράγουν ενέργεια στα ε, κράτη με χαμηλότερο εισόδημα της Ένωσης. Πώς θα διασφαλίσετε ότι δεν θα δώσουμε διπλές επιδοτήσεις στα εργοστάσια που παράγουν ηλεκτρισμό από άνθρακα. Εάν πρώτα απ' όλα τους δώσουμε δωρεάν δικαιώματα και μετά μέσω του Ταμείου Αντιστάθμισης δώσουμε και πάλι επιδοτήσεις, Δίνουμε δυο φορέ επιδοτήσει στον άνθρακα που παράγει ηλεκτρισμό. Θέλω λοιπόν να πει σαφώ η Επιτροπή ότι τα δωρεάν δικαιώματα και το Ταμείο Αντιστάθμισης δεν θα χρηματοδοτήσουν και τα δύο την παραγωγή ενέργεια από άνθρακα. Πρόεδρο ευχαριστώ. Η συνάδελφο Πεντιτσίνη για το EFDD. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε. Εδώ πέρα κάθομαι Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, σα ευχαριστώ πολύ. Μια ερώτηση όσον αφορά το νέο πρόγραμμα το οποίο προβλέπεται και βλέπουμε ότι έχουμε 32 33 εκατομμύρια ευρώ όσον αφορά τις διασυνδέσεις για τον τομέα των μεταφορών. Και προβλέπεται επίσης να γίνουν και επενδύσεις όσον αφορά την ενέργεια. Από τα 33,2 τα 5 δισεκατομμύρια προβλέπονται για τα δίκτυα ενέργειας ενώ 640 περίπου εκατομμύρια προβλέπονται για τις τρεις πρώτες μελέτες οι οποίες θα λάβουν χώρα και βλέπω ότι κυρίως χρηματοδοτούνται μελέτες. Οι μελέτες αυτές κοστίζουν 5 εκατομμύρια κάθε μία και προβλέπονται και άλλες μελέτες οι οποίες θα στοιχήσουν 10 εκατομμύρια ευρώ. Συνεπώς, θα ήθελα να γνωρίζω τι ακριβώς χρηματοδοτούμε μέσω των μελετών αυτών. Για ποιο λόγο κοστίζουν τόσο ακριβά αυτές οι μελέτες. Και επίσης, για να χρηματοδοτήσουμε όλες αυτές τις μελέτες, για ποιο λόγο χρειάζονται 70 περίπου δισεκατομμύρια ευρώ για το περίοδο μέχρι το 2020 και πραγματικά θα είναι αξιόπιστες μελέτες αυτές, θα έχουμε συγκεκριμένα υλοποιήσιμα πορίσματα. Σας ε, ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ όλους τους συναδέλφους για αυτόν τον πρώτο γύρο ερωτήσεων. Δίνω ευθύ αμέσω τον λόγο στον Επίτροπο για να απαντήσει στις ε, ερωτήσεις που υπέβαλαν οι συντονιστές. Έχετε το λόγο. Ε, Ευχαριστώ πολύ. Να απαντήσω <clears throat> πρώτα απ' όλα σε μία ερώτηση που, έγιναν, που έγινε από πολλούς και από τον κύριο Έκουτ και από τον κύριο Τόρβαλτς που αφορά την παρουσία μας στις ε, συναντήσεις κορυφής για την κλιματική αλλαγή όπως ξέρετε μία από τις δυνατότητε που έχουν οι αντιπρόεδροι είναι να καθορίζουν ποιος θα είναι παρόν στο Συμβούλιο, σε διεθνείς συναντήσεις, στο Κοινοβούλιο. Αυτό είναι αρμοδιότητα που ο Πρόεδρος ε, ανέθεσε στους αντιπροέδρους. Οπότε, Έχουμε βεβαίως ε, τις ε, συνήθεις ε, συναντήσεις μεταξύ επιτρόπων και του αντιπροέδρου που συντονίζει. Εκεί παίρνουμε αποφάσεις. Και η απόφαση που πήραμε είναι ότι στη Λίμα θα πάω εγώ. Εκεί για όλη τη βδομάδα της υπουργική ε, συνάντησης θα είμαι εγώ. Ως τακτικός εκπρόσωπος παράλληλα πάντα έχουμε επαφές σε όλα τα επίπεδα. Και ορισμένες φορές ο αντιπρόεδρος ε, είναι σε επαφή. Γιατί προσπαθούμε να έχουμε διπλωματικές επαφές σε κάθε επίπεδο για να επιτύχουμε στο Παρίσι Πρέπει να είμαστε σε επαφή με όλα τα έθνη των ΗΠΑ, με όλου του εμπλεκόμενου. Είναι τεράστιο καθήκον αυτό. Γι' αυτό ζητήσαμε να μα βοηθήσει και η κυρία Μογκερίνη. Γι' αυτό επιπλέον αξιοποιούμε και τα γραφεία εκπροσώπησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε 40 χώρες για να δείξουμε πόσο εμπλέκεται η Ένωση για να δούμε τις ανησυχίες των χωρών αυτών, τι θέλουν να επιτύχουν στη Λίμα και το Παρίσι και να προετοιμάσουμε το Παρίσι. Ήδη από τώρα συνεργαζόμεθα με την επερχόμενη Γαλλική Προεδρία, με τον μόνιμο πρέσβη για την κλιματική αλλαγή. Οπότε εργαζόμεθα σε όλα τα επίπεδα. Καταλαβαίνετε ότι αν επιτύχουμε μεγάλη επιτυχία στο Παρίσι, στην ε, τελετή υπογραφής θα θέλουν να πάνε πολύ. Εγώ θα εργαστώ πάρα πολύ μέχρι το Παρίσι, ούτω ώστε στο Παρίσι να έχουμε δεσμευτικούς στόχους. Να είστε λοιπόν σίγουροι ότι θα παρευρωθώ στη Λίμα, θα συνεχίσω να διαπραγματεύομαι με πολλές χώρες και τελικά θα αποφασίσουμε ποιος θα πάει στο Παρίσι. Αλλά ε, κάθε πράγμα στον καιρό του. Έχουμε εκπροσώπηση. Αλλά μη φοβηθείτε ότι δεν θα είμαστε αρκετά αποτελεσματικοί. Αν εργαστούν περισσότεροι θα επιτύχουν περισσότερο. Εγώ θα πάω στη Λίμα. Αλλά αν κάποιος ε, πρέπει παράλληλα κάποιος να έρθει σε επαφή με κάποιους στην Κίνα και τις ΗΠΑ θα υπάρξει συνεργασία. Αυτή είναι η αντιμετώπιση μας. Δεν έχει ληφθεί λοιπόν ε, μία απόφαση μία για πάντα. Ο αντιπρόεδρος αποφάσισε ότι εγώ θα πάω στη Λίμα, το δικό μου τηλέφωνο θα έχουν. Λοιπόν, άλλα θέματα τώρα. Ερωτήσει του κυρίου Μπέλετ. Για τη διαρροή άνθρακα. Σημαντικό θέμα που έχει απασχολήσει πολλούς. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο έχει αναφέρει τις αρχές ε, δωρεάν δικαιώματα και αυτά θα συνεχιστούν. Και η αρχή των δωρεάν δικαιωμάτων, όπως είπαν η ε, αρχή κρατών και κυβερνήσεων, πρέπει να δώσει σιγουριά στον κλάδο. Αλλά επίσης πρέπει να υπάρξει σφαιρική ανάλυση ούτω ώστε να καταλήξουμε σε νομοθετική πρόταση. Επίση, οι αρχή κρατών κυβερνήσεων πρέπει να υπάρχουν κριτήρια αναφορά για το πώ θα επιτύχουμε πρόοδο. Αυτό είναι θετικό. Αλλά πρέπει να το κάνουμε πιο λεπτομεριακό. Και επίση, σαφέ μήνυμα. Θέλουμε πιο αποτελεσματικέ εγκαταστάσει που δεν θα πρέπει να επιβαρυνθούν με νέο κόστο άνθρακα. Και αυτό είναι σαφέ. Όλα αυτά μαζί πρέπει να καταλήξουν σε διατύπωση νομοθεσίας, σε διάλογο με τους εταίρους. Πότε λοιπόν θα υποβληθεί αυτή η νομοθεσία. Αυτή είναι η πιο σημαντική ερώτηση. Θα προτιμούσα όσο δυνατόν νωρίτερα βέβαια. Αλλά κοιτάξτε, το θέμα της διαρροής άνθρακας δεν μπορεί να συνδεθεί με το θέμα του αποθυματικού σταθερότητας, γιατί αυτό το MSR είναι πολύ πιο προχωρημένο στην εξέτασή του. Άρα, δεν λέω ότι πρέπει να το περάσουμε με ταχεία διαδικασία, αλλά όσο το δυνατόν ταχύτερα να επιδιώξουμε έναν φιλόδοξο συμβιβασμό. Αυτό θέλει η Κομισιόν και ξέρουμε ότι μπορούμε να βασιστούμε και στη δική σας στήριξη. Αλλά δεν θα είναι εύκολο. Δεν θα είναι εύκολο. Διότι Ήταν δύσκολο να καταλήξουμε σε συμβασμό στο Συμβούλιο. Για ορισμένου δεν επαρκούν αυτοί οι συμβασμοί, αλλά ήταν δύσκολη η επίτευξή του, του συμβασμού αυτού. Καταλήξαμε σε κάτι που δεν ήταν αυτό που θέλαμε ω Κοινοβούλιο και Επιτροπή, αλλά παρόλα αυτά είναι φιλόδοξο στόχο που μπορούμε να τον παρουσιάσουμε στο Παρίσι. Ο Ματίας Γκρότε είπε ότι δεν καταλαβαίνουμε τι ακριβώς γίνεται με την πυρηνική ενέργεια και με τις ενεργοβόρες ε, εγκαταστάσεις στον τομέα της παραγωγής ενέργειας. Έχουμε, έχουμε σαφείς στόχους. Θέλουμε να είμαστε παγκόσμιοι ηγέτες στις ανανεώσιμες. Είμαστε περίπου στο 40% του ηλεκτρισμού μέσω ενέργειας. Αυτή τη στιγμή. Ενώ άλλες χώρες είναι πολύ πιο πίσω. Ποιο είναι το πρόβλημα τώρα για τη χρήση ανανεώσιμων. Ένα μεγάλο πρόβλημα. Ότι δεν έχουμε όλη εσωτερική αγορά ενέργειας. Έχουμε κλειστές εθνικές αλλαγές. Ε, αγορές, συγγνώμη. Οι διαμεθοριακές ε, δοσοληψίες είναι δυσχερείς. Ε, τα δίκτυα δεν είναι ευφυή. Οι κανόνες δεν είναι διαφανείς και σαφείς. Αν θέλουμε λοιπόν φιλόδοξους στόχους για τα ανανεώσιμα, Πρέπει να έχουμε μια πραγματική εσωτερική αγορά ηλεκτρισμού. Αυτό θα κάνει ο αντιπρόεδρος Σεύκοβιτς. Θέλει πρώτα απ' όλα μια φιλόδοξη μελέτη να κάνει ένωση με στόχο να υπάρξει πραγματική εσωτερική αγορά ενέργειας με διασυνδεδεμένα δίκτυα, με ανανεώσιμες. Γιατί υπάρχει πολύ περιθώριο στο νότο και στο βορρά, στη Βόρεια Θάλασσα Υπάρχουν τρομερές δυνατότητες παραγωγής ενέργειας. Το άλλο πρόβλημα που πρέπει να αντιμετωπίσουμε είναι η ενεργική ασφάλεια. Να διαφοροποιήσουμε τους προμηθευτές μας και τις πηγές μας και να καταλάβουμε ότι σε μερικές χώρες θα πρέπει να μειωθεί η παραγωγή από πυρηνικές ε, πηγές. Αυτό το απαιτεί και η Επιτροπή γιατί χρειαζόμαστε πολύ αυστηρές προδιαγραφές ασφάλειας. Ξεκινούμε το, τη δουλειά μας ταυτόχρονα σε διάφορα έργα. Μιλάμε για, το, για την πρόταση των 300 δισεκατομμυρίων και αυτή τη βδομάδα θα αρχίσουμε να εξετάζουμε το μελλοντικό πρόγραμμα της Κομισιόν. Αυτή τη βδομάδα δηλαδή θα το οριστικοποιήσουμε, τώρα το, το, το εξετάζουμε. Γι' αυτό δεν μπορώ να σας απαντήσω τώρα. Είμαστε στη διαδικασία αναθεώρησης όλων των προτάσεων που έχουν υποβληθεί και αξιολογώντας την ε, δυνατότητα που έχουν να προχωρήσουν σε, με βάση τα όσα έχουν συμβεί στο παρελθόν. Εμείς δεν θα βάλουμε προτάσεις στο πρόγραμμα που ξέρουμε ότι δεν πρόκειται να προχωρήσουν. Γιατί έχουμε πάρα πολλή δουλειά μπροστά μας και πρέπει να αναπτύξουμε όλες τις προτάσεις που σχετίζονται με το πλαίσιο του 2030 για το ETS, για τους τομείς εκτός ε, ε, ETS, για την οδηγία ενεργειακής αποδοτικότητας και η Κομισιόν παραμένει αφοσιωμένη στο να είναι πιο φιλόδεξη. Και αυτό αφορά και τους στόχους μας για την κλιματική αλλαγή. Είναι πολύ σημαντικό να έχουμε στο Παρίσι φιλόδοξους στόχους, γιατί έτσι θα έχουμε και μεγαλύτερη νομοποίηση για, στις διαπραγματεύσεις μας για την ενεργειακή αποδοτικότητα. Υπάρχει λοιπόν ένα περιθώριο κινήσεων που αφήνει τα συμπεράσματα του Συμβουλίου και η Κομισιόν εξακολουθεί να πιστεύει ότι η συνθήκη λέει πολύ ξεκάθαρα ποιες είναι οι πλειοψηφίε που απαιτούνται για τη λήψη αποφάσεων στην νομοθεσία. Κατανοούμε λοιπόν ότι το Συμβούλιο θέλει να έχει συνένεση σε αυτά τα ζητήματα, γιατί είναι σημαντικά, γιατί αφορούν την κλιματική αλλαγή, αλλά ταυτόχρονα θέλουν η ικανότητα της βιομηχανίας να, είναι, ε, να, είναι, να διατηρηθεί, οπότε η ισορροπία είναι σημαντικά, αλλά ε, θα πρέπει να διασφαλίσουμε ότι ακολουθούνται οι διατάξεις της συνθήκης που προβλέπουν την πλειοψηφία που χρειάζεται για την ε, λήψη αποφάσεων ε, στα θεσμικά όργανα. Είναι καλό λοιπόν το γεγονός ότι στο Συμβούλιο κάνουν προσπάθεια να ε, καταλήξουν σε συνένεση, αλλά ε, πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι η συνθήκη είναι σαφής. Δεν μας αποτρέπει από ε, το να υποβάλουμε νομοθετικές προτάσεις και να είμαστε φιλόδοξοι. Έχει ο καθένας το δικό του μερίδιο σε αυτή τη διαδικασία, το Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και θα προσπαθήσουμε να προωθήσουμε βεβαίως μια συμφωνία μεταξύ του Συμβουλίου και του Κοινοβουλίου με βάση τους πιο φιλόδοξους στόχους. Πάντω σε κάθε περίπτωση, όντα φιλόδοξοι, νομίζω ότι είμαστε στην ίδια ομάδα, είμαστε στην ίδια πλευρά και πρέπει να ε, επεξεργαστούμε έξυπνε στρατηγικές για να το πετύχουμε. Θα έχω λοιπόν ένα στενό διάλογο με τη δική σας επιτροπή για να δούμε πώς μπορούμε να προχωρήσουμε. Με εξέπληξε η ερώτηση του κυρίου Χωρίστη. Με με εξέπληξε όταν είπε ότι είμαι πεισμένο ότι η κλιματική αλλαγή είναι πραγματικότητα. Νομίζω ότι δεν θα βρείτε πουθενά αναφορά δική μου ότι δεν είναι πραγματικότητα κλιματική αλλαγή. Αν μελετήσετε αυτά που έκανα για την Τόχα, αυτά που είπα στη Βαρσοβία, θα διαπιστώσετε ότι είμαι πολιτικός που πιστεύει ότι η κλιματική αλλαγή η αλλαγή του κλίματος είναι πραγματικότης. Ότι τα αίτια της κλιματικής αλλαγής ουσοδός είναι ανθρωπογενή, ότι έχουμε τη δυνατότητα να αντιμετωπίσουμε τα λάθη και να διορθώσουμε τα λάθη που έχουμε κάνει και όσο ταχύτερα το κάνουμε τόσο λιγότερο θα μας κοστίσει στο μέλλον και πλέον πιστεύω ότι η πολιτική για την κλιματική αλλαγή μας δίνει δυνατότητα για ανάπτυξη, για απασχόληση, για ανάπτυξη τεχνολογιών, για πράσινες βιομηχανίες, για πράσινη ανάπτυξη, ότι δηλαδή υπάρχουν τεράστιες δυνατότητες. Ανήκα από τότε που ήμουν υπουργό Περιβάλλον στην πράσινη ομάδα, Green Group. Είμαι λοιπόν πολιτικός που πιστεύει ότι η πράσινη ανάπτυξη είναι πραγματικότητα και γι' αυτό πιστεύω ότι είναι σημαντικό να εργαστούμε σε αυτή την κατεύθυνση. Κυρίε και κύριοι, αυτό που θέλω να σας πω είναι ότι έχω τη βούληση να αντιμετωπίσω φιλόδοξα το θέμα της προώθησης του πακέτου 2030 για να επιτύχουμε στη Λίμα φιλόδοξους στόχους. Με ρωτήσατε τι θέλει να επιτύχει η Κομισιόν στη Λίμα. Θέλει να δημιουργήσουμε ένα σύστημα που να μας εγγυάται ότι όλα τα κράτη-μέλη θα έχουν συγκεκριμένους στόχους για την βελτίωση του κλίματος το πρώτο τρίμηνο του 2015. Ένα σύστημα σαφές επιτήρησης, ελέγχου, εξακρίβωσης για να δούμε ποιο είναι το επίπεδο αυτών των ε, δεσμεύσεων για να μπορέσουμε να τις συγκρίνουμε, να τις αθρήσουμε για να επιτύχουμε τη μείωση της αύξησης της ε, θερμοκρασίας ούτω ώστε να είναι λιγότερο από δύο βαθμοί και αν είναι ανεπαρκές αυτό, γιατί θα είναι ανεπαρκές, πρέπει να κάνουμε κατόπιν μία μεγαλύτερη προσπάθεια στο Παρίσι. Επίσης θα θέλαμε να έχουμε μία σαφή αντίληψη των βασικών τουλάχιστον αρχών του διαπραγματευτικού κειμένου που θα υποβληθεί στο Παρίσι για να επιτύχουμε αυτούς τους δεσμευτικούς στόχους. Αυτό θέλαμε. Θέλουμε να επιτύχουμε στη Λίμα και στο Παρίσι θα θέλουμε περισσότερα. Θα θέλαμε όλα τα κράτη του κόσμου, ανεπτυγμένα ή όχι, να θέσουν τους στόχους τους που να μας επιτρέψουν με δεσμευτικούς στόχους να μειώσουμε την αλλαγή του κλίματος εντός λογικών πλαισίων. Αλλά βήμα το βήμα όπως είπα και να μην ε, προτρέχουμε θεωρώντας ότι θα επιτύχουμε ή θα αποτύχουμε σε κάθε φάση. Η Λίμα είναι ένα βήμα, το Παρίσι θα είναι το επόμενο να εργαστούμε για να επιτύχουμε στη Λίμα και μετά θα έχουμε πολύ συγκεκριμένες διπλωματικές επαφές, πολύ έντονες, για να καταλήξουμε σε δεσμευτική συμφωνία στο Παρίσι που θα μας επιτρέψει να επιτύχουμε τους στόχους μας. Γιατί ένα είναι σαφέστατο. Το εξή. Η έκθεση των εμπειρογνωμόνων δεν αφήνει περιθώριο αμφιβολιών. Είναι μια έκθεση στην οποία συμμετείχε πολύ ενεργά η Ένωση. Χρηματοδότησε, αλλά συμμετείχε και με εμπειρογνώμονες και με ε, ένα τμήμα των ιδεών. Είναι λοιπόν ε, ουσιαστική έκθεση, έχει διανεμηθεί σε όλους ε, τους πολιτικούς που ασχολούνται με το θέμα αυτό, σε όλες τις χώρες του κόσμου και είναι προφανές ότι θέτει το πλαίσιο δράσης. Γι' αυτό πρέπει να εργαστούμε για να επιτύχουμε ικανοποιητικά αποτελέσματα στη, ρήμα, στη λίμα που να προπαρασκευάζουν το Παρίσι. Και ελπίζω να συνεργαστώ με την κοινοβουλευτική αντιπροσωπεία που θα μεταβεί στη Λίμα. Θέλω να είμαι σε μόνιμη επαφή με τον πρόεδρο και τα 12 μέλη που την αποτελούν. Με αυτόν τον τρόπο θα έχουμε μια ε, ευχερή ανταλλαγή απόψεων, ούτω ώστε να καταλήξουμε σε κοινή γραμμή προώθησης των θέσεών μας μέσω συνεργασίας. Σας ευχαριστούμε. Ας Ξεκινήσουμε τώρα τον δεύτερο γύρο παρεμβάσεων. Λάρα Ιούζο, ο πρώτος ομιλητής. Παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, και εγώ να σας καλωσορίσω στην Επιτροπή μας. Σας ευχαριστώ που ενώ αυτή τη βδομάδα έχετε τόσο πολλή δουλειά, ήρθατε εδώ και δηλώσατε ότι θέλετε να συνεργαστείτε διαφανώς με το Κοινοβούλιο. Αναφερθήκατε επανειλημμένα κατά την παρέμβασή σας στο σύστημα ITS. Ε αυτό το σύστημα διαμορφώθηκε ως ελεύθερη αγορά για να μειωθεί το κόστος της μείωσης των εκπομπών. Αλλά τι συνέβη. Ε, υιοθετήσαμε κάποιες νόρμες ad hoc, ορισμένες έχουν ε, ξεπεραστεί, είναι ξεπερασμένο και το σύστημα λοιπόν δεν ήταν τόσο απλό ούτε τόσο ευχερές όσο είχε θεωρηθεί. Θέλω να αφαιρθώ στις κρατικές ενισχύσεις που ε, ενέκρινε η προηγούμενη Επιτροπή για να αντιμετωπιστούν τα έμεσα στοιχεία κόστους του ETS που έχουν επίπτωση στην τιμή του ηλεκτρισμού. Αυτές οι κρατικές ενισχύσεις έγιναν στρέβλωση του ανταγωνισμού. Ξέρω ότι δεν είστε υπεύθυνο για τον ανταγωνισμό, αλλά ε, έχει μεγάλη επίδραση. Βέβαια, να ληφθούν μέτρα για να αποφύγουμε την μεταφορά εγκαταστάσεων σε τρίτες χώρες, αλλά πρέπει να αποφύγουμε επίσης τις τρευλώσεις στο εσωτερικό της αγοράς ενέργειας. Ερώτηση. Τι θεωρείτε για αυτό το μέτρο που πήρε η προηγούμενη Επιτροπή και τι μέτρα πιστεύετε ότι πρέπει να ληφθούν τώρα για να επιλύσουμε αυτά τα προβλήματα στρέβλος ανταγωνισμού που έχουμε αυτή τη στιγμή στην Ένωση. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ, ο Πρόεδρος προκειμένου να κινηθούν καλύτερα εργασίες μας. 13 έχουν ζητήσει το λόγο. Σας ζητώ λοιπόν, όπως έκανε και η κυρία Γιούζο, να περιορίσετε την παρέμβασή σας στο 1,5 λεπτό, προκειμένου να μπορέσουμε όλοι να μιλήσουμε. Ο κύριος Τζολάιν έχει το λόγο. Uh, Ευχαριστώ. Κύριε Επίτροπε και από τη δική, μας πλευρά, από τη δική μου πλευρά κάθε επιτυχία σας εύχομαι. Το Συμβούλιο αποφάσισε ότι οι στόχοι για τις ανανεώσιμες ε, και για την ανεργική ε, αποδοτικότητα δεν θα πρέπει να είναι δεσμευτικές. Εσείς τώρα πρέπει να ε, εφαρμόσετε αυτές τις κατευθύνσεις. Θα υπάρχουν αλλαγές, θα υπάρξουν αλλαγές στις οδηγίες, θα υπάρχει ένα άλλο σύστημα διακυβέρνησης. Δεύτερο, ε, ερώτημα. Στην ακρόαση είχατε, είχε αναφερθεί ότι αντέχεται να υπάρχει μια σύγκρουση ε, συμφερόντων. Ε, ως Επίτροπος για το κλίμα θα πρέπει να είστε ε, υπέρ του, των, ε, των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και φοβάμαι ότι ο μέσο ηλεκτροπαραγωγής ε, θα αποτελέσει εμπόδιο, εμπόδιο στην ε, ε, διάδοση των ανανεώσιμων. Εσείς πώς θα αντιμετωπίσετε αυτή την κατάσταση. Αυτό το, την, τα δύο συστήματα, το, το σύστημα δημοπράτησης και το σύστημα τροφοδότησης του δικτύου. Τι θα κάνετε με αυτά. Τρίτο ερώτημα. Αναφερθήκατε στις οδικές μεταφορές. Πολύ καλό. Έχουμε το πρόβλημα ότι η ενέργεια είναι πολύ φτηνή, Κάτι που σταματά την ανάπτυξη στα, των ηλεκτρικών ε, και των υβριδικών αυτοκινήτων. Τι θα κάνετε σε αυτό το τομέα. Κύριο Σπίακα έχει το λόγο. Το, το μικρόφωνο σας παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε. Όταν κοιτώ τα συμπεράσματα του Συμβουλίου, διαπιστώνω ότι υπάρχει μια διάσταση. Πώς, ε, ποια είναι η προσωπική σας άποψη για το σύστημα εμπορίας εκπομπών. Θα πρέπει οι τιμές να διαμορφώνονται από την αγορά ή όπως πρότεινε την τελευταία φορά το Κοινοβούλιο οι τιμές να αυξάνονται ε, μέσω διαφόρων νομοθετικών δραστηριοτήτων. Ποια είναι η δική σας η προσωπική άποψη σε σχέση με το ζήτημα αυτό. Η αγορά θα πρέπει να ορίζει τις ή θα πρέπει να ρυθμίζονται νομοθετικά. Το δεύτερο ερώτημα ε, είναι λεπτομερής, ε, είναι λεπτομεριακή. Είμαι από την Πολωνία και συγκεκριμένα στο 2.7 λέει στα συμπεράσματα το, το Συμβουλίο λέει ότι θα πρέπει να δημιουργηθεί ένα αποθεματικό 2%. Στην τέταρτη παύλα λέει ότι η απόφαση των κρατών μελών με συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Επενδυτικής Τράπεζας, Τράπεζας Επενδύσεων, θα, θα λαμβάνονται οι αποφάσεις και η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων έχει ακολουθήσει μια πολιτική που καθιστά πολύ δύσκολη την ε, πίστοση σε επενδύσεις, στον τομέα των επενδύσεων για τα πυρηνικά εργοστάσια. Τι θέλετε να κάνετε αυτό και τι ακριβώς εννοείτε με την, ε, ε, εννοείτε με την φράση με συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων. Ευχαριστώ κύριος ε, Φλόρενς. Ευχαριστώ. Μιλήσαμε πολύ για τη Λίμα και το Παρίσα και για τους, στόχους, τους του Κοινοβουλίου και για το αν θα είναι δεσμευτική ή όχι η στόχη, αλλά αυτό που με ενδιαφέρει εμένα είναι τι συμβαίνει με τα κράτη-μέλη εκείνα που δεν επέτυχαν τους στόχους τους για το 2020. Τι θέλετε να κάνετε με αυτούς. Η Ευρώπη μπορεί να έχει επιτύχει τους στόχους της, αλλά αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι κάποιοι δούλεψαν και κάποιοι δεν δούλεψαν. Και θα ήθελα να μου πείτε αν η κατάσταση αυτή μπορεί να συνεχιστεί. Εγώ στις ε, μικρομεσαίες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην εκλογική μου περιφέρεια θα αντιμετωπίσω πολλές δυσκολίες να τους το εξηγήσω. Ο κύριος Παρνιού, αντιπρόεδρος μας, έχει το λόγο. Κύριε Επίτροπε. Κύριε Επίτροπε, με ιδιαίτερη ευχαρίστηση ανταλλάσσουμε απόψεις μαζί σας εδώ στην Επιτροπή μας για πρώτη φορά λίγες εβδομάδες μετά τον δοριοσμό σας στη νέα σας αυτή θέση. Τρεις ερωτήσεις κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε. Μας είπατε πριν από λίγο ότι ο στόχος μας είναι να καταλήξουμε σε δεσμευτικούς αλλά λογικούς στόχους. Πρώτη ερώτηση λοιπόν. Το Πράσινο Ταμείο μέχρι στιγμής έχει 2,3 δισεκατομμύρια ευρώ και είναι όλα υποσχέσεις χρηματοδότησης, ενώ ξέρουμε ότι ο πραγματικός μας στόχος είναι μέχρι το 2020 να έχουμε φτάσει στα 100 δισεκατομμύρια δολάρια. Τα κράτη-μέλη έχουν συγκριμνοποιήσει την συνεισφορά τους στις 28 Οκτωβρίου του 2014 λογικά πρέπει να έχει γίνει κάτι τέτοιο. Δεύτερη ερώτηση. Ο Μπαράκ Ομπάμα, ο Αμερικανός Πρόεδρος, προβλέπει μια ημιδεσμευτική συμφωνία όσον αφορά την κλιματική αλλαγή, εν μέρη δηλαδή δεσμευτική. Βλέπουμε ότι ε, ήδη αντιμετωπίζουμε πάρα πολλές δυσκολίες από το γεγονός ότι το 2009 στην Κοπενχάγη δεν είχαμε δεσμευτική συμφωνία. Θα ήθελα λοιπόν να γνωρίζω αν εσείς έχετε ήδη μία συγκεκριμένη άποψη όσον αφορά την προσέγγιση αυτή των ΗΠΑ και μία εν μέρη δεσμευτική συμφωνία. Τρίτη ερώτηση. Η Κίνα γίνεται μία όλο και πιο ελκυστική χώρα όσον αφορά τις επενδύσεις σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αντίθετα, εμείς στην Ευρώπη δεν καταφέρνουμε να προσελκύσουμε ξένα κεφάλαια, ενώ βλέπουμε ότι οι αναδυόμενες οικονομίε προσελκύουν όλο και περισσότερα κεφάλαια επενδύσεων στις ανανεώσιμε πηγές ενέργειας. Ποια μέτρα προβλέπετε εσείς στην Ευρωπαϊκή Ένωση προκειμένου να καταφέρουμε να προσελκύσουμε κι εμεί ανάλογε επενδύσει. Σα ευχαριστούμε. Ο κύριο Φαρή έχει το λόγο. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Σας ευχαριστούμε πολύ κύριε Επίτροπε που ήρθατε στη δική μας την Επιτροπή σήμερα. Θα ήθελα να αφαιρθώ λίγο στην ενεργειακή απόδοση, στην ενεργειακή αποδοτικότητα. Νομίζω ότι λείπουν ακόμα πάρα πολλά δίκτυα διασυνδέσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και αυτό δεν μας βοηθά στο να πετύχουμε έναν βασικό μας στόχο, όσον αφορά δηλαδή την ενεργειακή απόδοση. Αν είχαμε για παράδειγμα το κατάλληλο επίπεδο ευρωπαϊκών διασυνδέσεων, τότε θα είμαστε σε θέση, για παράδειγμα, στην Ιβηρική Χερσόνησο να έχουμε πολύ χαμηλότερες ενεργειακές τιμές. Μιλήσαμε, αν δεν κάνω λάθος, τον Οκτώβριο για το ζήτημα αυτό, για την έλλειψη ευρωπαϊκών ενεργειακών διασυνδέσεων. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επίσης θα πρέπει να μας παρουσιάσει συγκεκριμένε προτάσεις χρηματοδότησης προκειμένου να υλοποιηθούν αυτά τα δίκτυα ενεργειακής διασύνδεσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά όσον αφορά το Connecting Europe Facility βλέπουμε ότι υπάρχει μια χρηματοδότηση πάρα πολύ χαμηλή. Και βλέπουμε ότι καλύπτονται χρηματοδοτικά μόνο κάποια έργα τα οποία δεν θα αποδώσουν οικονομικά. Θα ήθελα λοιπόν να γνωρίζω κύριε Επίτροπε ποια είναι τα νέα μέσα χρηματοδότησης τα οποία προβλέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προκειμένου να επιλύσει το πρόβλημα αυτό θα προβλεφθούν κάποια επιπλέον κονδύλια. Και στη συνέχεια, θεωρείτε εσείς ότι έχετε τα απαραίτητα μέσα όσον αφορά τα υφιστάμενα προβλήματα διασύνδεσης. Ευχαριστούμε πολύ. Η κυρία Ροντρίγκε Ρουμπί έχει το λόγο. Όπως ξέρετε, στην ομάδα μας μας απασχολεί ιδιαίτερα το θέμα του TTIP, και οι ενδεχόμενες επιπτώσεις του το περιβάλλον. Συγκεκριμένα να αναφερθώ σε ένα έγγραφο το οποίο διέρευσε τον Ιούλιο στη Washington Post όπου λέγεται ότι στο κεφάλαιο για την ενέργεια υπάρχει μια δεσμευτική ρήτρα με τις Ηνωμένε Πολιτείε που λέγεται ότι εγγυάται εξαγωγές πετρελαίου, εγγυώνται οι Ηνωμένε Πολιτείε εξαγωγές πετρελαίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πώς λοιπόν μπορούμε να αποφύγουμε αυτήν την οικονομική και περιβαλλοντική επιβάρυνση που σημαίνει η εισαγωγή ορυκτών καυσίμων από τις Ηνωμένες Πολιτείες και τον Καναδά και ποια είναι η γνώμη σας για την εισαγωγή αυτών των ε, ασφαλτούχων εδαφών από τον Καναδά, των ασφαλτούχων άμμων. Επίσης υπάρχει οδηγία για την ποιότητα των καυσίμων. Θα ήθελα να μου πείτε πώς μπορεί να συμβάλλει στη μείωση των ε, αερίων θερμοκηπίου. Ευχαριστώ πολύ. Ο Αντιπρόεδρος το λόγο. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε. Τρία ζητήματα θέλω να θίξω. Το πρώτο το ανέφεραν ήδη πολλοί συνάδελφοι. Πώς μπορούμε να καταφέρουμε να πετύχουμε τους μη δεσμευτικού στόχους στα πλαίσια του ETS και πώς θα πετύχουμε τελικά τους γενικότερους στόχους μας αν αυτοί δεν είναι δεσμευτικοί. Βλέπουμε ότι υπάρχουν πάρα πολλά κράτη-μέλη τα οποία τα οποία δεν πρόκειται να πετύχουν τους στόχους αυτούς, ακόμα και τους δεσμευτικούς στόχους. Προβλέπονται επιπλέον εγγύησεις λοιπόν επίτευξης αυτών των στόχων. Δεύτερον, υπάρχουν πάρα πολλέ στρατηγικέ στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και γενικότερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση όσον αφορά την κλιματική αλλαγή και όσον αφορά την ενέργεια. Μια στρατηγική όσον αφορά επίση την ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού. Αλλά δεν υπάρχει σαφή διασύνδεση ανάμεσα στην πληθώρα αυτή των στρατηγικών. Ποιο είναι το γενικότερο σχέδιο, ποιο είναι το γενικότερο πλαίσιο, αν θέλετε, στρατηγική μα όσον αφορά την κλιματική αλλαγή και την ενέργεια. Βλέπουμε ότι υπάρχουν πολλές διαφορετικές μορφές ενέργειας οι οποίες προωθούνται. Κάποιες από αυτές είναι επιζήμιες για το περιβάλλον, ενώ είναι ευνοϊκές για τις επιχειρήσεις. Ποια συγκεκριμένη στρατηγική μπορούμε λοιπόν να ακολουθήσουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ποιο είναι το γενικότερο στρατηγικό πλαίσιο. Τρίτο ζήτημα. Τα σχέδια κοινού συμφέροντος. Στη στρατηγική που μας παρουσιάσατε, το 90% των σχεδίων αυτών έχουν να κάνουν με τις εγκαταστάσεις φυσικού αερίου αυτή θα είναι η ευρωπαϊκή πολιτική όσον αφορά την ενέργεια, να αναλώσουμε τελικά όλα μας τα χρήματα, όλα μας τα κονδύλια στις εγκαταστάσεις φυσικού αερίου ή προβλέπετε να έχουμε και κάποιους νέους στόχους όσον αφορά την ενεργειακή αποδοτικότητα. Ευχαριστούμε. Το λόγο έχει η κυρία Εύη. Σας ευχαριστώ. Όσον αφορά το ETS, να επανέλθουμε στο ζήτημα αυτό, το προηγούμενο μήνα το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο είπε ότι θα πρέπει να μειώσουμε τις εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα 40% μέχρι το 2030. Αυτή τη στιγμή γίνονται διαπραγματεύσεις με την Ελβετία προκειμένου να συνδεθούμε με το δικό του σύστημα ETS. Και ο Γερμανός Υπουργός Περιβάλλοντος μας είπε ότι στο μέλλον το σύστημα ETS θα μπορούσε να συνδεθεί και με το κινέζικο σύστημα ETS. Πιστεύετε ότι θα είναι δυνατότητα διασύνδεση αυτή αν οι στόχοι που έχουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι καθαρά εγχώροι και εθνικοί. Και όσον αφορά την υλοποίηση επίσης του συστήματος αυτού. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έδωσε τη δυνατότητα στον Διεθνή Οργανισμό Πολιτικής Αεροπορίας να αναλάβει τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου να μειωθούν οι εκπομπές από τις αεροπορικές μεταφορές του 2016. Διαφορετικά ενδεχομένως η Ευρωπαϊκή Ένωση να πρέπει να λάβει συγκεκριμένα μέτρα, για παράδειγμα όσον αφορά όλες τις πτήσεις εκείνες οι οποίες εισέρχονται ή φεύγουν από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ότι θα πρέπει ενδεχομένω από το 2016 και μετά να ενταχθούν στο σύστημα ETS. Ε από το 1990 και μετά η αεροπορική κυκλοφορία έχει αυξηθεί και βλέπουμε ότι οι εκτιμήσεις του ΙΚΑΟ είναι ότι η κυκλοφορία των αεροπλάνων θα αυξηθεί, θα εξαπλασιαστεί στο μέλλον. Ποια μέτρα λοιπόν προβλέπετε εσείς όσον αφορά τις αεροπορικές μεταφορές και τις εκπομπές τους μέχρι το 2016. Η κυρία Σουίτσα έχει το λόγο. Ευχαριστώ. Να καλωσορίσω τον Επίτροπο Κανιέτε και τον ευχαριστώ που θεώρησε σωστό να έρθει να έχουμε αυτή την ανταλλαγή απόψεων έχουμε διαπιστώσει ότι υπάρχει ήδη. Βλέπουμε τι επιπτώσεις τη κλιματική αλλαγή. Πρέπει λοιπόν να την αντιμετωπίσουμε. Το είπατε κι εσείς. Η κλιματική πολιτική δεν μπορεί να λειτουργήσει αν δεν παίξει το ρόλο του και ο κλάδος, οι επιχειρήσεις. Και η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει βεβαίως ε, να θέτει τις καθεντήριε γραμμές παγκόσμια. Απαντήσατε σε κάποιες ερωτήσεις που ήθελα να θέσω, αλλά Πώς ε, στοχεύετε να παίξετε σωστά το ρόλο σας, ε, να το βάρος της Ένωσης να πείσει τις μεγάλες δυνάμεις και τις επιχειρήσεις να μειώσουν τις εκπομπές. Γιατί μέχρι στιγμής το έχουν αρνηθεί. Στην επιστολή του κυρίου Γιούγκερ λέει ότι θέλει να εστιάσετε στις ανανεώσιμες και ότι αναμένει να είμαστε ηγετική δύναμη στα θέματα αυτά και αναφέρεται και στη διαφοροποίηση των προμηθευτών και της οδούς εισαγωγών και θέλει επίσης να είστε ισχυρός διαπραγματευτής. Τι θα κάνετε για να επιτύχετε όλους αυτούς τους στόχους. Σεβόμενοι την κλιματική μας πολιτική. Και τώρα, μία ερώτηση για κάτι που με ενδιαφέρει ιδιαίτερα. Ξέρω ότι η Ενεργειακή Ένωση είναι αρμοδιότητα του κυρίου Σεύκοβιτς, αλλά θα ήθελα να μας πείτε ποια είναι η δική σας γνώμη για, για τον ε, αγωγό, αεραγωγό ε, της ε, Αδριατικής. Γκαρθία Πέρεθ. Ε, ευχαριστώ Πρόεδρε. Κάποιες ερωτήσεις που ήθελα να κάνω έχουν ήδη τεθεί από άλλους συναδέλφους, οπότε θα ασχοληθώ με ένα συγκεκριμένο θέμα. Ο σύντροφος μου, ο κύριος Γκρότε, αναφέρθηκε στο θέμα της πυρηνικής ενέργειας στην απάντησή σας, κύριε Επίτροπε, είπατε ότι υπάρχουν κάποια εμπόδια αυτή τη στιγμή για, την ανανεώση, για τις ανανεώσιμες και ότι πρέπει να τις προωθήσουμε περισσότερο, σύμφωνο, απόλυτα. Πρέπει οπωσδήποτε, να επιτύχουμε τους στόχους μας για τις ανανεώσιμες. Αλλά σε κάποιες περιπτώσεις είναι δύσκολο να επιτύχουμε το σωστό ενεργειακό μείγμα να αναπτύξουμε δηλαδή τις ανανεώσιμες εάν μείνουμε στην ε, πυρηνική ενέργεια. Έχουμε ένα κεντρικό σύστημα πυρηνικό που έληξε τώρα και που θέλουμε να παρατείνουμε μέχρι το 2030. Δηλαδή θα έχει ορισμένες εγκαταστάσεις μας θα έχουν 60 χρόνια ζωής ή το σύστημα καλύτερα. Και η ίδια η Κομισιόν είχε πει ότι δεν είχε λάβει ενημέρωση στα πλαίσια του άρθρου 37 της συνθήκης Ευρατόμ που θα της επέτρεπα, επέτρεπε να, ε, αξιο, να αξιολογήσει τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις ε, του πυρηνικού τομέα. Έχετε εσείς κύριε Κανιέτε πληροφόρηση. Λήφθηκε πληροφόρηση για τον τομέα αυτό. Γιατί είναι θέμα ασφάλειας. Είναι θέμα ασφάλειας και για τον κλάδο και για τους πολίτες που ζουν γύρω από αυτές τις πυρηνικές εγκαταστάσεις. Και δεν θα πρέπει λοιπόν να τεθεί εν αμφιβόλιο η ανάπτυξη του σωστού ενεργειακού μείγματο. Ευχαριστώ. Thank you, Chair. Um, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Όσον αφορά την αντιμετώπιση τη κλιματική αλλαγή, κύριε Επίτροπε, προφανώ μπορούμε να αλλάξουμε την νομοθεσία, αλλά πώ μπορούμε να αλλάξουμε την συμπεριφορά των ανθρώπων. Έχουμε την νομική, αν θέλετε, και την εθελούσια προσέγγιση και το πρόβλημα με την κλιματική αλλαγή είναι ότι χρειάζεται η συμβολή και των δύο στα πλαίσια τη νομοθεσία θα πρέπει να εξηγήσουμε στου πολίτε μα ω πολιτικοί για ποιο λόγο κάνουμε ό,τι κάνουμε, αλλά όσον αφορά τώρα την εθελούσια οδό, το πιο σημαντικό είναι να ενημερώσουμε του πολίτε μα προκειμένου να αλλάξουν συμπεριφορά. Πώ μπορούμε να ενημερώσουμε λοιπόν καλύτερα του πολίτε μα όσον αφορά το οικολογικό αποτύπωμα των προϊόντων που αγοράζουν προκειμένου να καταφέρουμε να πείσουμε τους πολίτες να αγοράζουν προϊόντα τα οποία παράγονται τοπικά. Καταλαβαίνετε ότι θα πρέπει να τους ενημερώσουμε για όλα αυτά τα ζητήματα και ενδεχομένω να πρέπει να συνδέσουμε το ζήτημα αυτό με το ζήτημα των μεταφορών που αναπτύξετε πριν από λίγο. Ευχαριστούμε. Ο κύριος Τζορίνιου έχει το λόγο. Σας ευχαριστώ κύριε Επίτροπε. Έχω ένα επιπλέον ερώτημα για τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για το πακέτο για το κλίμα εν ώψη 2030. Μία από τις αποφάσεις ήταν να οριστεί ένα στόχος 15% για τη δέσμευση. Έθεσε και ο συνάδελφος Σωρία ένα ερώτημα, δεν θα το επαναλάβω. Ρώτησε πώς ε, αυτή η δέσμευση μπορεί να χρηματοδοτηθεί από κοινού με τα έργα κοινού ενδιαφέροντος. Πώς θα εξασφαλιστεί η παρακολούθηση της επίτευξης του στόχου αυτού. Τι θα συμβεί σε μια χώρα η οποία σκοπίμως δεν συνεισφέρει στην επίτευξη του στόχου αυτού και ποιες είναι οι δυνατότητες που έχουν οι χώρες που θέλουν να επιτύχουν τους στόχους που έχουν τεθεί αλλά που εμποδίζονται γιατί πάντοτε το ζήτημα είναι να ε, υπάρχουν δύο ε, ε, μέρη σε αυτή τη συμφωνία. Ο κύριος Γραμματικάκης παρακαλώ. Χαίρομαι για την παρουσία του κυρίου Πιτρόπου εδώ και για την ενδιαφέρουσα συζήτηση. Εγώ θα επιμείνω μόνο σε μία ερώτηση δική μου, γιατί οι υπόλοιπε νομίζω ότι απαντήθηκαν με ικανοποιητικό καμιά φορά τρόπο και άλλοτε με θολό και αόριστο. Για μένα η εξοικονόμηση ενέργειας, ε, κύριε Πρόεδρε και κύριε Επίτροπε, είναι ένας κύριος περιβαλλοντικός στόχος κατά τους ειδικού και μένα που συμβαίνει να είμαι καθηγητής φυσικής. Δυστυχώς όμως γνωρίζετε ότι ο στόχος αυτός που είναι περίπου 1,5% ετησίως παραμένει ενδεικτικός και όχι δεσμευτικός. Αυτό επιτρέπει σε κάποιες ευρωπαϊκές κυβερνήσεις να τον παραμερίσουν ή να παρουσιάσουν πλαστά μέτρα για την εκπλήρωση του στόχου. Δυστυχώς ένα παράδειγμα είναι η χώρα μου, η Ελλάδα, που πρότεινε, συνεμπεριέλαβε την εξίσωση φόρου πετρελαίου κίνησης και θέρμανσης και επίσης την επέκταση του μετρό της Αθήνας και την κατασκευή του μετρό Θεσσαλονίκης για την εκπλήρωση του στόχου. Είναι φανερό ότι αυτά ίσως δεν ικανοποιούν τις οδηγίες. Θα ήθελα λοιπόν να ρωτήσω τον κύριο Επίτροπο επί τη βάση τριών σημαντικών λέξεων που είπε επιτήρηση, έλεγχος και εξακρίωση και το δεύτερο πώς θα διορθώσουμε τα λάθη μας να μου απαντήσει εάν μπορεί στο πώς πραγματικά ο στόχος αυτός του 1,5% θα γίνει δεσμευτικός και ουσιαστικός. Ευχαριστούμε ο κύριος έχει το λόγο. Κύριε Επίτροπε, πριν από λίγο σας έκανα μια ερώτηση, αλλά δυστυχώς δεν έλαβα απάντηση. Επομένως, θέτω εκ νέου την ερώτησή μου αυτή πιο σύντομα αυτή τη φορά. Αναφέρομαι στο νέο πρόγραμμα Ευρωπαϊκών Διασυνδέσεων. Το πρόγραμμα αυτό δέχθηκε χρηματοδότηση 33 δισεκατομμυρίων ευρώ όσον αφορά τις διασυνδέσεις μεταφορών, τη διασυνδέση στην πληροφορική και τις διασυνδέσεις στον τομέα της ενέργειας. Για να χρηματοδοτούν όμως όλα αυτά τα προγράμματα χρειάζονται περίπου 70 δισεκατομμύρια ευρώ. Ποιες ιδιωτικές επενδύσεις μπορούν να γίνουν που θα είναι αξιόπιστες επίσης. Και επίση, ποιε εγγύσει έχουμε ότι δεν θα σπαταληθούν τα χρήματα αυτά σε μια περίοδο οικονομική κρίση. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. κυρία Ρίκοζη έχει το λόγο. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Δύο ερωτήσεις, κύριε Επίτροπε. Πρώτον, αναφερθήκατε στις επενδύσεις των 300 δισεκατομμυρίων ευρώ για τρία χρόνια ως Επίτροπος για το κλίμα και την ενέργεια. Ποιες συγκεκριμένε προτάσεις έχετε να κάνετε σε σχέση με αυτό το επενδυτικό σχέδιο. Γιατί είπατε ότι θα το συζητήσουμε τις επερχόμενες εβδομάδες. Οι δικές σας οι απόψεις ποιες είναι όσον αφορά αυτό το επενδυτικό σχέδιο. Δεύτερον, μετά τα συμπεράσματα του Συμβουλίου στι 23 και 24 Οκτωβρίου, θεωρώ ότι υπάρχει μια φράση στο 2.7 που είναι κάπω προβληματική, που λέγεται ότι χρειάζεται ένα αποθεματικό προκειμένου να αυξηθεί η ενεργειακή αποδοτικότητα και να εξυγχρονιστούν τα ενεργειακά συστήματα των κρατών μελών. Τι σημαίνει εξυγχρονισμό των ενεργειακών συστημάτων κρατών μελών θα εξυγχρονίσουμε τις μονάδες παραγωγής ηλεκτρισμού από άνθρακα, θα εξυγχρονίσουμε τις μονάδες παραγωγής που χρησιμοποιούν ορυκτά καύσιμα. Τι εννοούμε με τον όρο εξυγχρονισμό. Ευχαριστούμε. Ο κύριος Ντάνς, τελευταία ερώτηση παρακαλώ. Uh, Κάτι πολύ σύντομο και για τους συναδέλφους σας, αλλά ίσως και εσείς ε, μπορείτε να μας ε, φωτίσετε λιγάκι. Είπατε ότι όταν αποφασίσατε τις, τις προτεραιότητές σας θα εξετάζατε και προτάσεις που θα μπορούσαν να έχουν μια κρίσιμη μάζα υποστήριξης. Πώς θα πάρετε αυτές τις αποφάσεις. Θα ρωτήσετε και το Κοινοβούλιο. Πώς θα μας διαβολευτείτε για να δείτε τι είναι εφικτό και τι όχι. Γιατί για τα θέματα αυτά το τι είναι εφικτό ή όχι δεν συμπίπτουν όλες οι απόψεις. Ευχαριστούμε. Νομίζω ότι υποβάλαμε πάρα πολλές ερωτήσεις στον Επίτροπο. Έχετε περίπου 10 λεπτά κύριε Επίτροπε για να απαντήσετε σε όλες τις ερωτήσεις. Κοιτάξτε, από κοινού απαντήσει σε κάποιες ερωτήσεις, καθότι υπάρχουν πάρα πολλές ερωτήσεις οι οποίες ομοιάζουν μία με την άλλη, μπορείτε να απαντήσετε συλλογικά σε κάποιες ερωτήσεις. Κυρία Γιούσου, για το θέμα των κρατικών ισχύσεων, τι θα κάνω. Ο υπεύθυνο ε, Επίτροπος θα αναλύσει και θα δει κατά πόσο είναι συμβατές. Κύριε Λάινεν, Κάνατε πολλές ερωτήσεις. Αλλά κυρίως μιλήσατε για την ενεργειακή αποδοτικότητα και είπατε ότι δεν είναι δεσμευτικό. Αλλά είναι σαφές αυτό. Τόσο η Επιτροπή όσο ο πρόεδρος δηλαδή και εγώ θα επιμένουμε ότι χρειάζεται τουλάχιστον σε ευρωπαϊκό επίπεδο δεσμευτικό στόχος και μετά η διακυβέρνηση θα πρέπει να μας ε, επιτρέψει να προσπαθήσουμε να εξηγήσουμε σε όλους ότι όλα τα κράτη πρέπει να κάνουν προσπάθεια, αλλά χρειάζεται ευελιξία. Γιατί δεν είναι στην ίδια κατάσταση όλα τα κράτη-μέλη. Δεν μπορούν να εφαρμόσουν τα ίδια μέτρα ενεργειακής αποδοτικότητας, ούτε με την ίδια ένταση. Διότι τα σημεία κίνηση είναι διαφορετικά. Πολύ διαφορετικά. Και αυτό είναι σαφές. Για μένα τουλάχιστον. Για τις ανανεώσιμες. Βεβαίως τι εμπόδια αντιμετωπίζουμε για να τις προωθήσουμε. Οι ανανεώσιμε έχουν τρία προβλήματα. Πρώτον, η καινοτομία. Πρέπει να αναπτύξουμε ανανεώσιμες ενέργειες, αλλά και ενέργειες για την αποθήκευση τη ενέργεια. Πρέπει λοιπόν να κάνουμε πολλές επενδύσεις όσον αφορά την αποθήκευση στις τεχνολογίε για να επιτρέψουμε τη χρήση των ανανεώσιμων. Δεύτερον, Το δεύτερο πρόβλημα είναι ότι οι αγορές δεν είναι διασυνδεδεμένες. Πρέπει λοιπόν να ενισχύσουμε την διασύνδεση και τα έξυπνα δίκτυα για να διευκολύνουμε τις ε, μεταφορές τις διασυνοριακές. Αυτό είναι θεμελιώδες. Αν καταφέρουμε να επιτύχουμε αυτήν την εσωτερική αγορά θα αναπτύξουμε και τις άλλες, ε, και ε, και τις άλλες πλευρές. Αυτό είναι σαφές. Και μετά είχα και μια ερώτηση από τον κύριο Πατσά για το ποια είναι η άποψή μου για το ETS. Το σύστημα ETS θα πρέπει να είναι προσανατολισμένο στην αγορά. Μπορούμε να εφαρμόσουμε ένα αποθεματικό για να ε, αποφύγουμε τις ε, διακοιμάνσεις, αλλά αυτό δεν, είναι, δεν, δεν πρέπει με πολιτικές αποφάσεις να ορίζονται οι τιμές θα πρέπει να ε, μπορούμε εμείς ε, με βάση τα δικαιώματα να επηρεάζουμε τα πράγματα αλλά δεν πρέπει να επηρεάζουμε τις τιμές. Το πρόβλημα δεν είναι, τον δεν είναι πρόβλημα υψηλών τιμών, είναι το να δώσουμε ε, σήμα στις οικονομίες ότι οι επενδύσεις κατευθύνονται στις τεχνολογίες χαμηλού άνθρακα. Τώρα, ποια είναι το πρόβλημα με τη σύνδεση θα πρέπει να υπάρχει κάποια ομοιογενής ε, σύγκριση. Ε, συνεργαζόμαστε με τους Ελβετούς αυτόν τον καιρό και δεν έχουμε λύσει ακόμα όλα μας τα προβλήματα, αλλά θα είναι καλό να συνδέσουμε την ελβετική αγορά με τη δική μας αγορά. Αν ε, στο μέλλον αναπτυχθούν και άλλες αγορές με βάση τους ίδιους προσανατολισμούς, τότε καλύτερα. Τότε θα είναι ακόμα καλύτερα τα πράγματα. Το όνειρό μας θα ήταν δηλαδή να ε, ε, δημιουργήσουμε μια παγκόσμια αγορά. Ρωτήσατε, ποια είναι η συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Απενδύσεων. Και επανέρχομαι στο νέο πακέτο που σχετίζονται με το πακέτο Juncker. Ο πρόεδρος θα προτείνει ένα πακέτο 300 δισεκατομμυρίων για τις επενδύσεις και, την απασχόληση. Ένας από τους τομείς στους οποίους υπάρχουν ανάγκες για περισσότερες επενδύσεις είναι ο τομέας της ενέργειας. Διότι οι επενδύσεις που απαιτούνται στον συγκεκριμένο τομέα ανέρχονται σε 204, 204 δισεκατομμύρια το χρόνο για την ηλεκτροπαραγωγή. Σημαίνει αυτό ανανεώσιμες για την βελτίωση των δικτύων που είναι απαρχαιωμένα και αναποτελεσματικά σε πολλές χώρες και η αντικατάσταση αυτών των δικτύων με έξυπνα δίκτυα για την ενεργειακή αποδοτικότητα των κτηρίων. Εκεί χρειαζόμαστε τεράστια ποσά στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την ενεργειακή αποδοτικότητα στη βιομηχανία. αυτό μπορεί πραγματικά να ε, απαιτήσει μεγάλο μέρος του πακέτου Juncker και εγώ κάνω ό,τι περνά από το χέρι μου για να περάσουν κονδύλια στον εξυγχρονισμό του δικτύου, την ενεργειακή αποδοτικότητα των κτηρίων και της βιομηχανίας. Αν δείτε όλα τα έργα που εκτελούνται, τα κοινού ενδιαφέροντος που βρίσκονται υπό επεξεργασία υπάρχουν πάρα πολύ μεγάλες ευκαιρίες. Τι μπορούμε να κάνουμε. Έχει συσταθεί μια ομάδα και συνεργαζόμαστε με την Τράπεζα Επενδύσεων για το πώς μπορούμε να γίνουμε πιο αποτελεσματικοί ώστε να ε, συγκεντρώσουμε και ιδιωτικές επενδύσεις, όχι μόνο μέσω των παραδοσιακών δάνειων, αλλά και μέσω άλλων χρηματοδοτικών εργαλείων που μπορούν να ε, μας αποφέρουν ε, περισσότερα κεφάλαια. Ερώτηση για το τι γίνεται με τις χώρες που δεν ε, επιτυχάνουν τους στόχους. Έχουμε την οδηγία για την ενεργειακή αποδοτικότητα που λέει τι γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις και θα πρέπει να την εφαρμόσουμε. Στο νέο σύστημα που θα θέλαμε να είναι δεσμευτικό και φιλόδοξο θα πρέπει να δημιουργήσουμε ένα νέο σύστημα διακυβέρνησης και θα συζητήσουμε με το Κοινοβούλιο ποιος θα είναι ο καλύτερος τρόπος για να το διαμορφώσουμε. Υπήρξε και ένα ερώτημα. Ο κύριος Παρνιών. Που ρώτησε τι συμβαίνει με την... Ποια είναι η κατάσταση με τις ΙΠΑ. Ε, το πρόβλημα είναι ότι ο πρόεδρος και το Κογκρέσο αυτή τη στιγμή έχουν διαφορετικές απόψεις και προκειμένου να ε, επιτύχουμε συμφωνία στο Παρίσι θα πρέπει να ε, εγκριθεί η στάση των ΗΠΑ από το Κογκρέσο όπως και εμείς θα πρέπει να εγκρίνουμε αυτό που θα κάνουμε και οι Αμερικανοί διαπραγματευτές θα πρέπει να βρουν έναν τρόπο ώστε να μπορούν με να κάνουν πράγματα αλλά ε, να διαμορφώσουν και με έναν έξυπνο τρόπο την νομοθετική ε, πράξη. Οπότε θα πρέπει να κάνουμε πάρα πολύ δουλειά με τους ε, νομικούς μας, γιατί το σημαντικό που θέλουμε εμείς να επιτύχουμε είναι να αναλυθούν δράσεις. Ο κύριος Φαρία μίλησε για, την, για τις διασυνδέσεις στην Πορτογαλία, το είπαν και άλλοι, είναι πάρα πολύ, είναι ξεκάθαρο. Ε, η Βαλτική, η Βυρική Χερσόνησο και τα νησιά είναι, ε, αντιμετωπίζουν προβλήματα με τη διασύνδεση και ο συμβιβασμό στον οποίο ε, καταλήξαμε είναι το 10% που μπορεί σίγουρα και 15% στο 2030. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στο 1,4% στην Ιβυρική Χερσόνησο. Αν ε, Ε, εφαρμόσουμε το, τον στόχο που θέλουμε ε, θα είναι 2,4% Και αυτή τη στιγμή εκπονούμε οικονομικές μελέτες για το αν είναι βιώσιμη ε, αυτή η προοπτική. Βασιζόμαστε στη συνεργασία των κρατών μελών. Αλλά αν θέλουμε να εργαστούμε προς μια πραγματική εσωτερική αγορά θα χρειαστεί να ενισχύσουμε τη διασύνδεση. Αλλά σε κάθε περίπτωση δεν θα είναι εύκολο το έργο αυτό. Ροντρίγκε. Είπε ότι υπάρχουν προβλήματα με την, ε, με την ενέργεια. Οπωσδήποτε η, συνθήκη αυτή το TTIP είναι σε φάση πολύ προκαταρκτική αλλά η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει μεγάλο συμφέρον σε πρόσβαση στην αγορά της Βόρειας Αμερικής για να διαφοροποιήσει τις πηγές της, ιδιαίτερα το φυσικό αέριο των ΗΠΑ. Κοιτάξτε κυρία Ροντρίγκε, η τιμή του φυσικού αερίου είναι τρεις ή τέσσερις ε, φορές υψηλότερη από ότι το φυσικό αέριο που έχει η βιομηχανία στο, ε, στις Ηνωμένες Πολιτείες και το ίδιο ισχύει και για την Κίνα. Συζητάμε με τους, Ρούσους, με τους Ρώσους ούτως ή άλλως για το δικό τους αέριο. Γι' αυτό λοιπόν το φυσικό αέριο που από τα ορυκτά καύσιμα είναι ας το πούμε έτσι λιγότερο μολύνων ρηπαίνων από τα άλλα μας είναι χρήσιμο για να διαφοροποιήσουμε τις πηγές ε, προμήθειας. Το έχει πει η Κομισιόν. Έχουμε αναφερθεί στα προβλήματα ενεργικής ασφάλειας. Οπωσδήποτε λοιπόν θα ήταν σκόπιμο να έχουμε πρόσβαση στο φυσικό αέριο και για λόγους ασφάλειας και για λόγους μείωσης ε, του κόστους ενέργειας να στηρίξουμε δηλαδή τις βιομηχανίες μας. Καταλαβαίνω τις ανησυχίες σας για αυτές τις ε, ασφαλτούχες ε, άμμους το, από τον Καναδά. Αλλά έχουμε ένα ποσοστό χρήσης τους. Και στα πλαίσια αυτού του ποσοστού μπορούμε να πάρουμε από που να είναι αυτές τις ε, ε, άμμους. Ο κύριος ε, Σάμπορ έθεσε το θέμα των στόχων για το 2020 και το 27% σε επίπεδο ενωσιακό. Τουλάχιστον έχουμε έναν ε, ενωσιακό στόχο. Και μετά με το σύστημα διακυβέρνησης θα πρέπει να διαμορφώσουμε τους μηχανισμούς. Πολλές φορές δεν ε, σκεφτόμαστε μηχανισμούς κυρώσεων. Είναι μηχανισμοί στήριξης πρέπει να σκεφτούμε πώς μπορούμε να αναπτύξουμε τις ανανεώσιμες σε όλες τις χώρες. Να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα για την εφαρμογή. Να υποστηρίξουμε δηλαδή τα κράτη-μέλη, να διευκολύνουμε το έργο των κρατών μελών, όχι απλώς κυρώσεις δηλαδή. Ο κύριος Πεντιτσίνη στη συνέχεια αναφέρθηκε στη χρηματοδότηση συγκεκριμένων ερευνών και προγραμμάτων. Ναι, ισχύει ότι οι πόροι που έχουμε για τα προγράμματα συνδέοντας στην Ευρώπη δεν επαρκούν, αλλά το πακέτο Juncker μας δίνει μια μεγάλη ευκαιρία για να ε, πιέσουμε γκάζι, για να πατήσουμε γκάζι στον τομέα αυτό. Και έχουμε λοιπόν προγράμματα πολύ πιο φιλόδοξα. Νομίζω ότι με αυτό ε, προσπάθησα να απαντήσω στις περισσότερες ερωτήσεις. Α, με συγχωρείτε. Α, η κυρία Ιράτσε. Δεν έχω τα στοιχεία αυτή τη στιγμή. Θα τα βρω και θα σας τα στείλω. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστούμε. Εξ ονόματος όλων θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Επίτροπο Αρία Κανιέτε για την διαθεσιμότητά του, για αυτή την ανταλλαγή απόψεων, για το ότι κατάφερε επίσης να απαντήσει συγκεκριμένα σε όλες τις ερωτήσεις που κατέθεσαν οι συνάδελφοι. Ολοκληρώνοντας αυτό το σημείο η συνεδρίασή μας. Η επόμενη συνεδρίαση της Επιτροπής μας θα λάβει χώρα στις 24 Νοεμβρίου. Πρόκειται για έκτακτη συνεδρίαση που θα γίνει από τις 7 το βράδυ στο Στρασβούργο και η επόμενη τακτική μας συνεδρίαση θα γίνει στις 3 και 4 Δεκεμβρίου στις Βρυξέλλες. Σας ευχαριστώ πολύ και όσοι ε, πρέπει να αποχωρήσετε αυτή τη στιγμή, σας παρακαλώ πολύ μην κάνετε θόρυβο και φύγετε σύντομα έτσι ώστε να ξεκινήσει και η συνεδρία των συντονιστών.